Äh, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να κηρύξω την έναρξη τη κοινή συνεδρίαση και εκ μέρου του συναδέλφου κ. Νταζόν και Äh, και του κυρίου Αλέκας να σας ε, χαιρετήσω θερμά όλους και να σας καλωσορίσω στην αίθουσα όπου θα συζητήσουμε κυρίως ε, θέματα αμυντικής, πολιτικής και ασφάλειας. Καλωσορίζω α, και τον κύριο Ολέκα. Ναι. Τον Υπουργό Άμυνας της Λιθουανίας. Ε, τα θέματα μας είναι εξαιρετικού ενδιαφέροντος δεδομένου είχαμε και την διακοινοβουλευτική συνεδρίαση, διυπουργική συνεδρίαση στο Βίλνιο πριν από μερικές εβδομάδες και αναμένουν τις, ε, την ενημέρωση και τα τελευταία δεδομένα όλα τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών. Ε, κύριε Ντονζόν, αναμένουμε μία επιτυχή συνεδρίαση και συνεργασία με το Συμβούλιο. Θα ήθελα να αναφέρω μερικά θέματα ε, τα οποία θέλουμε να συζητήσουμε. Καταρχάς θέλουμε ένα δικό χάρτη για μία εις βάθος ε, ε, και διαρθρωτική και ολοκληρωμένη συνεργασία. Αυτός είναι ο στόχος και της προσδοκόμενης λευκής βίβλου. Επίσης, ε, θέλουμε τη συνεργασία των, των άλλων συνδεδεμένων ομάδων σε θέματα κοινά ασφάλειας, άμυνας και βιομηχανικής ικανότητας, βιομηχανικών δυνατοτήτων συμμετοχής ε, σε αυτούς τους τομείς. Δεν είναι μόνο καθαρά οικονομικό ή χρηματοδοτικό το θέμα, αλλά είναι και πολιτικό το θέμα που έχει να κάνει με την εθνική κυριαρχία. Επίσης πρέπει να ε, πούμε ότι η Κομισιόν έχει υποβάλει μια πολύ ενδιαφέρουσα ε, ανακοίνωση σε αυτό το θέμα. Κύριε Υπουργέ, θεωρούμε την κοινή αυτή συναντήση με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων μεγάλη σημασία, διότι εάν η ευρωπαϊκή κοινότητα δεν ενισχύσει περισσότερο τη συνέργεια ε, σε τα θέματα της, ε, πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους ευρύτατους στόχους προστασίας και διαφύλαξης των συνόρων. 70% των Ευρωπαίων πολιτών σε όλα τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι χρειάζεται απόλυτα η ευρωπαϊκή ελοκλήρωση για, ειδικά για τον τομέα της ε, άμυνας. Άρα λοιπόν έχουμε ένα βαρύ έργο μπροστά μας και ανακαλύψουμε τα κοινά και να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Και ε, εσείς ως Προεδρεύων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πιστεύω ότι θα μας ε, εμπλουτίσετε με πληροφορίες και παρατηρήσεις τις οποίες θα μπορέσουμε να σημειώσουμε και να λάβουμε υπόψη στην έκθεσή μας η οποία έκθεσή μας ε, θα αναφέρει, ε, μια, θα, προβάλλει μια εις ανάλυση των δύο τομέων, ασφάλειας και άμυνας. Και θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον συνάδελφο κύριο Ντεζάν. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε εδώ σήμερα. Θα είμαι πολύ σύντομος. Πρώτα απ' όλα για το Υπουργό ξέρω ότι πρέπει να έρθει στις 4 ακριβώς, οπότε πρέπει να προλάβουμε, να έχουμε καρποφόρα συζήτηση μαζί του. Και ο Έλμαρ, από τη δικιά του πλευρά, συνόψισε πάρα πολύ καλά το τι διακυδεύεται για το Κοινοβούλιο στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Εννοείται ότι έχουμε κάποιες ανησυχίες, γιατί πολλά είναι τα ζητήματα, ίσως υπερβολικά πολλά. Και φοβούμεθα ότι η αυθονία των θεμάτων και των τομέων τελικά μπορεί να καταλήξει σε όχι πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις, παρόλο που βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή και πιστεύουμε εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι ήρθε πια η ώρα να συνειδητοποιήσουμε τις προκλήσεις που συλλογικά πρέπει να αντιμετωπίσουμε στον τομέα τη άμυνα. Θα μα τα πείτε κι εσείς. Απλώς να σα πω ότι για τη Πρώτα απ' όλα, στη διάσκεψη την διακοινοβουλευτική που ήταν αφιερωμένη στην πολιτική ασφάλεια και άμυνα το Σεπτέμβριο, μα υποδεχτήκατε τόσο καλά. Ήταν βέβαια στα πλαίσια, μάλλον παράλληλα με το Κίμνηστο Συμβούλιο που έλαβε χώρα. Με το ΝΑΤΟ μπορέσαμε λοιπόν να έχουμε πολύ ενδιαφέρουσε συζητήσει. Η διάσκεψή σα οργανώθηκε πραγματικά πάρα πολύ καλά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπήθηκε καλά πάλι, πράγμα που δεν συμβαίνει πάντα και από τα εθνικά κοινοβούλια. Εμείς δείχνουμε έτσι το ενδιαφέρον μας και καλά κάνουμε. Επίσης θέλω να αναφέρω εδώ και την παρουσία και το ενδιαφέρον της Λιθουανίας όσον αφορά τις ευρωπαϊκές αποστολές στα πλαίσια ακριβώς της μη στρατιωτικής δυνατότητας σχεδιασμού και διεξαγωγής επιχειρήσεων στο Μαλί, για παράδειγμα, και στο Κωσυφοπέδιο που είχαμε παλιότερα. Θα σας ακούσουμε. Είχαμε το θάνατο ενός τελωνιακού Λιθουανού στο βόρειο Κωσυφοπέδιο το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, τα συλληπιτήρια μας γι' αυτό. Κάτι το οποίο βέβαια δείχνει ότι καμία αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και αν είναι μη στρατιωτική, καμία δεν είναι χωρίς κίνδυνο. Πολλές φορές ακούμε κριτική για τις μη στρατιωτικέ αυτές τις αποστολές, ότι ίσως είναι πολύ επιφανειακές, ότι δεν είναι αρκετά φιλόδοξε. Ε, λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο επαγγελματισμό και η δέσμευση που αναλαμβάνουν όλοι επί τόπου είναι κάτι που πρέπει να υπενθυμίζουμε συνέχεια. Καμία δεν είναι χωρίς ε, κινδύνους. Πάντα είναι θέμα ασφάλειας και δυστυχώς είδαμε τι έγινε στο Κωσυφοπέδιο το Σεπτέμβριο. Συνεπώς, τα συλληπιτήριά μας στην Λιθουανία και στα μέλη της Λιθουανίας, είτε του στρατιωτικούς είτε του θελωνιακούς που συμμετέχουν στην αποστολή αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την υποδοχή που με επιφυλάξατε. Κύριε Ντονζά, κύριε Μπροκ, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, αξιότιμοι προσκεκλημένοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Πραγματικά με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι εδώ σήμερα και απευθύνομαι έτσι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω της Υποπιτροπής αυτής Ασφάλειας και Άμυνας. Είναι η πρώτη φορά που έχω την ευκαιρία να απευθυνθώ σε εσά και γι' αυτό και σας ευχαριστώ όλους ιδιαίτερος για την ευκαιρία που μου δίνετε να μοιραστώ μαζί σας τις ιδέες μου όσον αφορά την κατάσταση ασφάλειας και άμυνας στην Ευρώπη. Έχω εργαστεί στο Κοινοβούλιο εδώ και πολλά χρόνια. Ήμουνα και στην Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας, οπότε ειλικρινά νιώθω εδώ μεταξύ συναδέλφων. Είχα την ευκαιρία επίσης να συναντήσω πολλούς από εσά στο Βίλνιους στην διάσκεψη, την διακοινοβουλευτική για την ασφάλεια και την άμυνα, στην οποία αναφέρθηκε και ο Πρόεδρος. Εκεί είχαμε υψηλού επίπεδου συζητήσεις ουσίας. Οι οργανωτές ελπίζω να σας έδωσαν την ευκαιρία όχι μόνο να συζητήσετε, αλλά να ανακαλύψετε και το Βίλνιους ή να επισκεφτείτε και κάποιες άλλες πόλεις της Λιθουανίας. Ελπίζω να φύγατε με καλές εντυπώσεις από το Βίλνιους και ελπίζω να επιστρέψετε. Το εξάμεινο αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Λιθουανία και για την κυβέρνηση της Λιθουανίας αλλά και για όλους τους πολίτες. Η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα από τα θέματα για τα οποία συμφωνούμε 100% με την αντιπολίτευση. Και ομολογώ ότι δεν υπάρχουν πολλά τέτοια θέματα πάνω στα οποία να συμφωνούμε έτσι. Η Προεδρία λοιπόν για μας αποτελεί μια πρόκληση, μια πρόκληση και για τον δημόσιο τομέα μας. Αλλά να ξέρετε ότι κανένας οργανισμός, κανείς ε, δεν ε, ε, περιόρισε τις προσπάθειές του. Καθένα άλλο όλοι κάνανε όσο μπορούσαν περισσότερες προσπάθειες για να προχωρήσει η εμπειρία αυτή θετικά για όλους. Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι η Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επηρεάσει τη Λιθουανία και στο μέλλον και όλους τους θεσμούς της Λιθουανίας. Από την άλλη μεριά, ελπίζω ότι η Ευρώπη από τη δικιά της πλευρά θα γνωρίσει καλύτερα τη Λιθουανία έτσι μετά την Προεδρία μας. Ότι θα έχετε μάθει περισσότερα πράγματα για την ιστορία μας κατά τη λήξη του εξαμήνου αυτού. Είμαι αισιόδοξο και ελπίζω ότι το μέλλον θα είναι θετικό και για μας. Θέλω να αναφερθώ λιγάκι τώρα στους στόχους της Λιθουανικής Προεδρίας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας και να σας εξηγήσω ποιες είναι οι προσπάθειες της Λιθουανίας για την εφαρμογή της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Τους πρώτους μήνες της Προεδρίας είχαμε διάφορα εκδηλώσεις στο Βίλνιους και διάφορες συναντήσεις, σεμινάρια στη Γαλλία, στο Παρίσι. Μετά την ε, σημερινή συνάντηση πάμε στο Λονδίνο, όπου θα συζητήσουμε εκεί για το μέλλον των ομάδων μάχης. Όλα αυτά είναι θέματα με τα οποία η Λιθουανική Προεδρία θέλει να προχωρήσει τα θέματα της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και να τα προωθήσει στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Επίσης θέλω να σας αναφέρω ότι η Λιθουανία δεν έχει μόνο την Προεδρία, δραστηριοποιείται επίσης ενεργά περισσότερο από ποτέ στον τομέα της ΚΕΠΑ. Υπάρχουν 120 στρατιώτες Λιθουανοί στις ε, μονάδες αυτές μάχης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Λετωνία, τις κατοχώρες και τη Σουηδία. Επίσης, εκπαιδευτές στρατιωτικοί Λιθουανοί έχουν ε, συμμετάσχει στην εκπαιδευτική αποστολή στο Μαλί. Επίσης, προσφέρουμε και σκάφη στην ε, Αταλάντα για να διασφαλιστεί η ανθρωπιστική βοήθεια από τα Ηνωμένα Έθνη. Έτσι λοιπόν την Προεδρία δεν τη βλέπουμε μόνο σαν μια ευκαιρία για νέες πολιτικές προαιρότητες αλλά και σαν υποχρεώση να συμμετέχουμε ενεργά στην εφαρμογή των ήδη συμφωνημένων πολιτικών. Πάντα είναι ευχάριστο να μιλάει κανείς για τα επιτεύγματα. Όμως ξέρετε πολύ καλά ότι τον τελευταίο καιρό η Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα είναι πράγματα που συζητιούνται μάλλον με απεσιόδοξο πνεύμα. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει όλο και περισσότερες προκλήσεις ασφάλειας. Οι δαπάνες για την άμυνα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες μειώνεται. Συγχρόνως υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους πόρους που απαιτούνται και στους πόρους που είναι διαθέσιμοι και το κενό αυτό καλύπτεται από λόγια, πρωτοβουλίες που έχουν περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα. Κάτι το οποίο βέβαια δεν μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση. Υπό το φως της κρίσης, ο τομέας της άμυνας στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχει υποφέρει από τη λιτότητα. Ακόμα και εκεί που υπάρχει κάποια ανάκαμψη στην οικονομία, οι ευκαιρίες για αύξηση του προπολογισμού άμυνας είναι πολύ περιορισμένες. Τώρα θα σας πω δύο λόγια όσον αφορά τη χρηματοδότηση της άμυνας. Πιστεύω ότι τις στρατιωτικές μας ικανότητες και την ανάκαμψη της βιομηχανίας άμυνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα την καταφέρουμε μόνο όταν θα αλλάξει αυτή η τάση που υπάρχει όσον αφορά τις δαπάνες στην άμυνα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας, οι δαπάνες αυτές έπεσαν κατά 10% από το 2005 μέχρι το 2010 και από ό,τι φαίνεται άλλο 10% έπεσαν από το 2010 στο 2013. Με άλλα λόγια δηλαδή, τα τελευταία χρόνια η πτώση αυτή στις δαπάνες που πάνε στην άμυνα είναι κάτι το οποίο επιταχύνεται. Η διαδικασία αυτή καταλαβαίνετε ότι θα έχει τεράστιες συνέπειες, όχι μόνο στην ευρωπαϊκή βιομηχανία άμυνα, αλλά και όσον αφορά την θέση της ίδια τη Ευρώπης στον κόσμο. Δεν υπάρχει τρόπος να το ξεχάσουμε αυτό. συνεπώ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σημασία στο θέμα αυτό των αμυντικών δαπανών. Αυτές τις μέρες οι ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα και η Λιθουανία, αναφέρονται στην ανάπτυξη στρατιωτικών ικανοτήτων. Όμω, περισσότερο μιλάμε για την διαχείριση της μείωσης των δαπανών. Τον Δεκέμβριο οι ηγέτες κατώ και κυβερνήσεων θα πρέπει να ανακοινώσουν φιλόδοξα σχέδια και πρωτοβουλίες. Ακριβώς αυτό είναι που έχω υπόψη μου όταν σας έλεγα νωρίτερα ότι στην Ευρώπη υπάρχει μια πρακτική ρητορική και πρωτοβουλίων συμβολικών προκειμένου να καλυφθεί το κενό ανάμεσα στα χρήματα που απαιτούνται και στα χρήματα που είναι διαθέσιμα. Πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Για παράδειγμα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας δείχνει ότι οι ένοπλες δυνάμες είναι από τους οργανούς εκείνους που καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια στις χώρες μας. Άρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πιο καλές τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας ή οχήματα τα οποία να χρησιμοποιούν λιγότερα καύσιμα. Και τα χρήματα που θα εξοικονομήσουμε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κατάρτιση ε, στρατιωτικών, για παράδειγμα. Επίσης θα μπορούσαμε να επενδύσουμε τα χρήματα αυτά γενικότερα στην σαφιωτική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να, μια άλλη δουλειά για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας. Η αναθεώρηση αυτή πρέπει όντως να ξεκινήσει το Δεκέμβριο με το Συμβούλιο. Το Δεκέμβριο έχουμε τη δέκατη επέτειο της στρατηγικής αυτής. Πολύ συχνά σε τέτοιες συναντήσεις έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε αναθεώρηση. Όμως δεν είναι αυτό το πιο σημαντικό και εδώ θα σας παραθέσω δύο προτάσεις που αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή αυτή στρατηγική ασφάλειας. Λέει ότι η Ευρώπη ποτέ δεν ήταν τόσο ευημερούσα, τόσο ασφαλής και τόσο ελεύθερη η βία που συναντήσαμε, που απαντήσαμε μάλλον στις αρχές του 20ου αιώνα, τώρα έχει δώσει τη θέση της σε μια περίοδο ειρήνης και σταθερότητας. Μπορεί κανείς σήμερα να υποστηρίξει ότι τα λόγια αυτά ισχύουν ακόμα ή ότι είναι μια βάση για τη σημερινή Ευρώπη. Δεν νομίζω. Τα τελευταία δέκα χρόνια ο κόσμος γύρω από την Ευρώπη έγινε λιγότερο ασφαλής, περισσότερο ασταθής και πιο ριζοσπαστικός. Συγχρόνω, η ίδια η Ευρώπη από την πλευρά τη κλείστηκε πιο πολύ στον εαυτό της. Πολιτικά είναι λιγότερο φιλόδοξη και στρατιωτικά δεν είναι τόσο πολύ σε θέση να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις ακόμα και κοντά στα σύνορά της. Στα πλαίσια λοιπόν της αναθεώρησης της στρατηγικής αυτής θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι στο μέλλον οι Ευρωπαίοι πολίτες θα βρεθούν εκτεθειμένοι περισσότερο στην ανασφάλεια στις γειτονές χώρες. Αλλά επιπλέον πρέπει να θυμόμαστε ότι οι Ηνωμένε οι οποίες μέχρι τώρα ε, χρησιμοποιούσαν δυνάμεις στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν αποφασίσει όλο και περισσότερο να επικεντρώνονται σε άλλα σημεία του κόσμου και λιγότερο στην Ευρώπη. Συνεπώς η Ευρώπη πρέπει να ξανασκεφτεί ποιο είναι ο παγκόσμιος ρόλος της και κυρίως ποιο είναι ο ρόλος των στρατιωτικών της δυνάμεων στα πλαίσια της ευρωπαϊκής αυτής στρατηγικής ασφάλειας. Θέλω επίση να αναφέρω και νέες αναδιόμενες ε, απειλές, όπως είναι θέματα κυβερνοχώρου και ενέργειας. Πράγματα τα οποία δεν αναφέρονται στην σημερινή ευρωπαϊκή ε, στρατηγική ασφάλειας. Είναι όμως πολύ σημαντικά στοιχεία για μας και τις γείτονες χώρες. Ίσως θα ακούσατε ότι πρόσφατα υπάρχει το κέντρο αριστείας του ΝΑΤΟ για την άμυνα στον κυβερνοχώρο στο Ταλίν. Όπως επίσης υπάρχει και ένα κέντρο ενεργειακής ασφάλειας στο Βίλνιος που ξεκίνησε φέτος να λειτουργεί. Πολύ σημαντικά αυτά για να αντιμετωπιστούν οι αυξηνόμενες απειλές στην ε, περιοχή μας. Τώρα, το κύριο μήνυμά μου είναι ότι υπό το φως των αλλαγών που λαμβάνουν χώρα τα τελευταία χρόνια, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τώρα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο και να ενημερώσει το έγγραφο αυτό της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας. Έρχομαι τώρα στο θέμα των ε, εταίρων μας στα θέματα ασφάλειας. Μετά τις αμυντικές δαπάνες και την αναθεώρηση δηλαδή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας, που είπαμε ότι ελπίζουμε να αναθεωρηθεί τον Δεκέμβριο, έρχομαι στο θέμα των ε, εταίρων μας, στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Όπως ξέρετε, μια από τις κύριες προτεραιότητες της Λιθουανικής Προεδρίας είναι η ενίσχυση της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Ελπίζουμε ότι η διάσκεψη, η σχετική που θα λάβει η χώρα τον επόμενο μήνα στο Βίλνιους, θα καταλήξει στην υπογραφή αυτής της πολύ σημαντικής συμφωνίας σύνδεσης με την Ουκρανία και ελπίζουμε να μονογραφηθεί επίσης και αντίστοιχη συμφωνία με τη Γεωργία και τη Μολδοβία. Είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με τους εταίρους μας, τα ανατολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι τώρα οι συμφωνίες ε, που έχουμε αυτές δηλαδή οι σύνδεσεις δεν αναφέρουν τόσο τα θέματα της ασφάλειας και της άμυνας. Όμως είναι πολύ σημαντικό η Ουκρανία για παράδειγμα να μπει μέσα στην ευρωπαϊκή διαδικασία ολοκλήρωσης. Είναι μια γεωπολιτική αλλαγή η οποία θα αλλάξει το πρόσωπο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στους ανατολικούς της γείτονες. Από την άλλη μεριά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εκμεταλλεύεται πλήρως τις δυνατότητες που έχουν οι εταίροι στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Δεν υπάρχει τακτικός διάλογος ασφάλειας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους γειτονές της και όσο μάλλον ε, συνεργασία στρατιωτική σε διάφορα προγράμματα. Προσπάθειες που έγιναν μέχρι τώρα έχουν αποτύχει, έχουν γίνει ελάχιστε. Για παράδειγμα, οι χώρε μέλη θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνουν εκπροσώπου των χωρών εταίρων μα στι δυνάμει που αναπτύσσουν στα πλαίσια των διαφόρων επιχειρήσεών του με ελάχιστο ή καθόλου κόστο. Είναι κάτι το οποίο κάνει το ΝΑΤΟ και έχει αποβεί ιδιαίτερα αποφελέ. Γενικά μιλώντα λοιπόν, έχουμε παραδείγματα και με την Ουκρανία σε αποστολές του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν. Η σχέσεις μας λοιπόν με τους εταίρους μας στις αυτοτικές δραστηριότητες είναι κάτι που θεωρούμε ότι δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Θεωρούμε ότι δεν αποτελούν μέρος των πολιτικών μας με τους γειτονές μας. Και όταν υπάρχει τέτοια συνεργασία συμβαίνει μόνο σε ad hoc βάση δυστυχώς. Έτσι δεν αποφελούμαστε αρκετά από τις ικανότητες των γειτόνων μας. Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα έχουμε μια χώρα εταίρο και μια χώρα μέλος που μπορούν να προσφέρουν τις ίδιες δυνάμεις ανάπτυξης για μια ε, αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάντα προτιμάμε την ευρωπαϊκή χώρα. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι εταίροι μας από τρίτες χώρες τελικά δεν έχουν σχεδόν ποτέ την ευκαιρία να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις δικές μας, παρά μόνο εάν οι 28 ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούν να προσφέρουν τέτοιες ικανότητες. Και όπως καταλαβαίνετε, 20, όταν 28 ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούν να προσφέρουν αυτό που χρειάζεται μια επιχείρηση, ε, πόσο μάλλον θα δεν θα μπορούν άλλες τρίτες χώρες. Άρα λοιπόν Πώ είναι δυνατόν χώρε όπω η Γεωργία, η Μολδοβία, οι οποίε θα θέλουν να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκέ επιχειρήσει, πώ είναι δυνατόν τελικά να συμμετέχουν, έχουν την ικανότητα να το κάνουν αυτό. Προφανώ και δεν θα το έχουν. Γι' αυτό ίσω θα πρέπει εδώ να ισχύσει η αρχή τη θετική διάκριση. Δηλαδή να στηρίζουμε του εταίρου μα κάθε φορά που μπορούν να προσφέρουν κάποιε ικανότητε να τι δεχόμαστε. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η χρήση υπηρεσιών τις οποίες πληρώνουμε σε ιδιωτικές υπηρεσίες αν εμείς δεν έχουμε τις δυνατότητες να καλύψουμε τις ανάγκες. Έτσι, για παράδειγμα, η εκπαιδευτική αποστολή στο Μαλί πρόσφατα νίκιασε ελικόπτερα για την ε, Υγειονομική Εκένωση 5 εκατομμύρια για 6 μήνες. Του χρόνου θα πληρώσουμε πάνω από 10 εκατομμύρια για τις ίδιες αυτές υπηρεσίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως δεν απευθύνθηκε ποτέ στους εταίρους της να τους ρωτήσει αν μπορούν εκείνοι να βοηθήσουν και να δώσουν πιο φτηνά, με καλύτερους όρους τέλο πάντων αντίστοιχο υλικό. Συνεπώς, στην Προεδρία μας εμείς υπογραμμίζουμε τη σημασία που έχει η συνεργασία με τους εταίρους μας και ιδιαίτερα με τους γειτονές μας. Τέτοια συνεργασία είναι ε, ένας στόχος που πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί έτσι καλύτερα διαγράφει το περιβάλλον ασφάλειάς της. Με άλλα λόγια, η επένδυση στην ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας είναι μια καλή επένδυση σε στιγμές λιτότητας. Έρχομαι τώρα στις νέες αναδυόμενες προκλήσεις. Το πεδίο αυτό που θα ήθελα να συζητήσει σε βάθος το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο οποίο αναφέρθηκα πριν μιλώντας για την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας, είναι ακριβώς οι αναδιόμενες προκλήσεις ασφάλειας. Θα έλεγα ότι πρέπει να αλλάξουμε, να μην τις λέμε αναδιόμενες, γιατί τις έχουμε την τελευταία δεκαετία. Αλλά δεν έχουμε βρει καμιά καλύτερη περιγραφή από ό,τι φαίνεται. Ξάλλου μην ξεχνάμε ότι η Λιθουανία και άλλες χώρες που μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 εξακολουθούμε να τις αποκαλούμε νέες χώρες μέλη παρόλο που μετά από την ε, ένταξή τους δύο φορές υπήρξε διεύρυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν μιλάμε λοιπόν για αναδυόμενες προκλήσεις ασφάλειας συνήθως μιλάμε για τον κυβερνοχώρο και για θέματα ενέργειας. Εννοείται ότι είναι πολύ περίπλοκα τα θέματα αυτά. Αυτό σημαίνει ότι και η απάντηση που θα δώσουμε θα είναι επίση περίπλοκη. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μα τους κανόνες, τα στάνταρτ, τις επενδύσεις που θα κάνουμε, την ενεργό διπλωματία, τις αποτρεπτικές προσπάθειες κλπ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη δικιά της πραγματογνωμοσύνη είναι σε καλύτερη θέση από οποιοδήποτε άλλο να αναλάβει ηγετικό ρόλο για τέτοια μη στρατιωτικά θέματα όπως είναι οι απειλές στον κυβερνοχώρο και η ενεργειακή ανασφάλεια. Φυσικά, προβλήματα αυτού του είδους δεν μπορούν να λυθούν παρά μόνο σε στενή συνεργασία με άλλες χώρες και οργανισμούς, το ΝΑΤΟ πρώτα απ' όλα, και έτσι να υπάρξει συνεργασία και σε κέντρο όπως αυτό το κέντρο εργαστίας στο Βίλνιους και στο Ταλίν. Ελπίζω ότι με αυτό το πεδίο θα ασχοληθεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Θέλω να τελειώσω με μια αισιόδοξη κάπως νότα. Στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας η Ευρώπη είναι ικανή να κάνει περισσότερα από όσα νομίζει ότι μπορεί. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Η απεσιοδοξία είναι κολλητική. Είναι ήδη να ξεχνάμε ότι μέχρι πρόσφατα είχαμε 50.000 στρατεύματα από ευρωπαϊκές χώρες που είχαν αναπτυχθεί στο Αφγανιστάν. Από το 2005 μέχρι το φθινόπωρο φέτος αυτή η μικρή χώρα, η Λιθουανία, ηγήθηκε της ομάδας περιφερειακής ανοικοδόμησης στο Αφγανιστάν με ειδικέ επιχειρησιακές μονάδες. Το 2011, ευρωπαϊκές χώρες ήταν υπεύθυνε για να φέρουν σε πέρα τις περισσότερες αποστολές μάχης κατά την δράση του ΝΑΤΟ στη Λιβύη. Φέτος έχουμε την επιχείρηση Σερβάλ στο Μαλί, όπου η Γαλλία μόνη της ε, κατάφερε τόσα πολλά. Δεν είναι μυστικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τα καταφέρνει συχνά να αποφασίσει για κοινέ δράσεις. Αυτό οφείλεται σε έλλειψη πολιτικής βούλησης. Αύριο θα συζητήσουμε ένα από αυτά τα θέματα στο Λονδίνο. Η συζήτησή μας επικεντρωθεί στις ομάδες μάχης δεν έχουμε καταφέρει να τις αναπτύξουμε ενώ τις έχουμε εκπαιδεύσει. Έχει νόημα να συνεχίσουμε να τις κρατάμε. Οι ομάδες αυτές μάχης έχουν ε, συγκριθεί συχνά με το κανόνι στη Μόσχα του Τσάρου, το οποίο ενώ απ' έξω έδειχνε τόσο τέλειο δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Είναι όμω σαφέ από τα παραδείγματα που σα έδωσα μέχρι τώρα και είμαι πεπισμένο ότι όταν είναι κρίσιμη η κατάσταση τότε οι ευρωπαϊκέ χώρε μέλη και οι ένοπλε δυνάμεις μπορούν να δράσουν γρήγορα και αποτελεσματικά. Και θέλω εδώ να προσθέσω ότι πιστεύω ότι είναι ακόμα ικανέ γιατί μπορεί να χάσουν την ικανότητα αυτή στο μέλλον εφόσον δεν χρησιμοποιούνται. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το Δεκέμβριο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δώσει νέα όθηση και να δώσει ένα θετικό μήνυμα για την χρήση τους. Η Λιθουανική Προεδρία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για να τεθούν όλα αυτά σε εφαρμογή. Και πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι η δικιά σας Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας θα στηρίξει ενεργά τα κράτη-μέλη σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Θέλω να σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και την υπομονή σας. Επειδή έχουμε λίγο χρόνο, θα ξέρετε ότι θα απαντήσω σε μερικέ ερωτήσει, αλλά μην ξεχνάτε ότι πρέπει να πάρουμε το τρένο για το Λονδίνο σε λίγο και δυστυχώ ο χρόνο, η υπαλλήρια και τα τρένα δεν περιμένουν κανέναν άνθρωπο, ούτε καν τον Υπουργό Άμυνα. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Είστε εξαιρετικά πιστικός, θα έλεγα, και αποφασισμένος. Είναι αυτονόητο, το έχουμε πει πολλές φορές σε αυτήν εδώ την Επιτροπή, ότι μας ενδιαφέρει και υποστηρίζουμε η πολιτική και τα θέματα που αναφέρεται, Σκέφτομαι ιδιαίτερα την αναθεώρηση, την ανανέωση, την επικαιροποίηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας όπως αναφέρατε. Εδώ στα δικά μας ψηφίσματα μιλάμε για λευκή βίβλο θα πρέπει να ξεκινήσει ως μεθοδολογία αυτή η Λευκή Βίβλος χωρίς να περιμένουμε να μας παράσχει το Συμβούλιο μια έτοιμη Λευκή Βίβλο με το κλειδί στο χέρι. Ελπίζουμε όμως ότι αυτό το Συμβούλιο θα αποτελεί την αφετηρία για μια διαδικασία που θα αποσκοπεί στον καθορισμό προτεραιοτήτων της Ευρώπης, στην κατάρτιση των απειλών, των απειλών που θεωρεί ότι έχουν προτεραιότητα για την ασφαλειά της, και βάσει αυτής της διαπίστωσης ε, ελπίζουμε ότι θα μπορέσει έτσι να καταρτήσει μια πραγματική στρατηγική. Το επαναλαμβάνουμε διαρκώ στα εγγραφά μας. Ε, Πρόσεξε ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται την πολιτική γειτονία και το γεγονό ότι η κοινή πολιτική ασφαλείας και Άμυνα ε, θα έπρεπε πράγματι να αποτελέσει μία από τις διαστάσεις αυτής της πολιτικής γειτονίας διότι με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης όπως και της Νότιας ε, υπάρχουν σημεία σύγκληση σε θέματα ασφάλειας και άμυνας και πόροι οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από κοινού. Το θέμα αυτό είναι πολύ ευαίσθητο αλλά ε, και δεν μπορούμε φυσικά να το διαπραγματευτούμε εύκολα αλλά σίγουρα υπάρχουν σημεία συμμετοχής της επιχειρήσης μας που έχουν ενδιαφέρον να μελετήσουμε στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Για παράδειγμα νομίζω στο Αφγανιστάν ε, ε, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορούν να μας εμπνεύσουν για το ευρωπαϊκό μοντέλο. Το λόγο έχει ο κύριος Κάλλερ. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ Υπουργέ. Πράγματι σας αναγνωρίζω την έντονη δέσμευση της Λιουθανικής Προεδρίας ειδικά σε αυτό το θέμα και ήδη υποδείξατε τη συνεδρίαση στο Βίλνιος και πιστεύω ότι είναι σωστό να υποστηρίξουμε αυτήν την Προεδρία ιδιαίτερα και πολιτικά διότι αυτή τη στιγμή την χάνεται μία κάπως ε, μη φιλικής ε, μεταχείρισης από τις γειτονικές χώρες, από μερικές γειτονικές χώρες. Γι' αυτό λοιπόν εγώ ενθέρμω σας ευχαριστώ για την ε, υποστήριξή σας. Οπωσδήποτε από το 2005 στην Ευρώπη μέχρι το 2013 έχουμε 20% περικοπές του προϋπολογισμού. Αυτό είναι ένα γεγονός, όμως δεν είναι διόλου η σωστή απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Έχουμε εκφράσει τις επικριτικές μας απόψεις. Είπατε ότι θα υπάρξει μια σχετική ανακοίνωση. Το θέμα είναι ότι καλώς έχουν οι ανακοινώσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υλοποιούνται. Εδώ έχουμε ήδη συγκεκριμένα συμπεράσματα και πιστεύω ότι θα μπορέσετε στην διάσκεψη κορυφής να εφαρμόσετε μια στρατηγική από τα ψηλά στα χαμηλότερα έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε από το ύψιστο επίπεδο σε συγκεκριμένες αποφάσεις και να υπάρξει ένα θετικό, θετικά συμπεράσματα αυτής της ε, διάσκεψης. Επίσης όσον αφορά τις ομάδες Battle Πιστεύετε ότι θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε με μια νέα προσέγγιση ε, για τις ομάδες αυτές ή νομίζετε ότι θα υπάρξει μια νέα εντολή για την επεξεργασία μιας προσέγγισης σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας για πρώτη φορά ακούω αυτές τις ε, απόψεις από την πλευρά του Συμβουλίου ότι ενδεχομένως ε, αυτή θα είναι η πρόθεση ε, τη δέκατη μέρα του έτους ότι είναι μια καλή μέρα για να ξεκινήσουμε. Οποιαδήποτε μέρα είναι καλή για μας ε, για να ξεκινήσει κάτι σωστό. Όσον αφορά τώρα τη χρηματοδότηση και για το μηχανισμό ε, Αθήνα, Ατένα. Έγινε μια ανασκόπηση τακτική και θέλουμε να εντάξουμε ορισμένου μηχανισμούς στο πλαίσιο του Ατένα, ε, παραδείγματο χάρη δυναμικό, ανάπτυξη δυναμικού και ορισμένα άλλα στοιχεία. Τι συμβαίνει τώρα στο, τις διαβουλεύσεις που γίνονται μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Θα, θα αναθεωρηθεί αυτός ο μηχανισμός ώστε να εντάξει περισσότερα στοιχεία ή όχι. Αυτά κύριε Υπουργέ προς το παρόν. Ευχαριστώ. Θα ακούσουμε όλες τις ερωτήσεις, κύριε Πασκής. Εκτός μικροφόνου. Παρακαλώ, εκτός μικρόφωνο. Ε, θα ήθελα να μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό για την παρουσίασή του. Μας περιέγραψε πολλά προβλήματα και παρουσίασε και πολλές προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές θα χρειαστεί να καταλήξουν κάποια ανταπόκριση. Αναφέρθηκε στη συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους και το να δοθεί προτεραιότητα σε αυτή τη συνεργασία. Έχει η Λιθουανία παραδείγματα όπου εμείς χρησιμεύσαμε ως παράδειγμα. Επίσης θα ήθελα να μιλήσω για τη συνοδοκορυφή του Δεκεμβρίου στο Βίλνιου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κύριε Υπουργέ πέραν των νέων απειλών στις οποίες εκτιθέμεθα και που είναι αρκετά σημαντικές θα επικεντρωθείτε καθόλου στις παλιές απειλές ε, που ζει η Ευρώπη και ο κόσμος ε, τον τελευταίο καιρό αλλά για τις οποίες δεν έχουν γίνει πολλά όπως για παράδειγμα η κλιματική αλλαγή θα δώσετε καθόλου προσοχή σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Λίζακ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Σε λίγο θα αναχωρήσετε για το Λονδίνο. Ήθελα λοιπόν να σας κάνω μια ερώτηση όσον αφορά τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου. Όσον αφορά την κοινή πολιτική ασφαλής και άμυνας. ερώτηση μου είναι πολύ απλή. Θεωρείτε ότι ότι σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο αντιτεθεί στην ανάπτυξη της κοινή πολιτικής ε, άμυνας και ασφαλείας ούτως ή άλλως το Ηνωμένο Βασίλειο αντιτίθεται στο να γίνει σε αυτή η πολιτική θεωρείτε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο. Όλες οι χώρες οι οποίες επιθυμούν την εμβάθυνση της κοινή πολιτικής ε, άμυνας και ασφάλειας, αυτές οι χώρες θα πρέπει να συνεχίσουν προ αυτή την κατεύθυνση ακόμα και αν εκφράσει την αντίθεση του Ηνωμένου Βασίλειου. Η δεύτερη μου ερώτηση αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι εταίροι μα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι Αμερικανοί εταίροι μας ε, υπογραμμίζουν εδώ και μήνες ότι η μείωση του αμυντικού προπολογισμού επηρεάζει αρνητικά τις ικανότητες άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τις δυνατότητες μας δράσης σε επιχειρήσεις εκτός της Επίρου μας. Θα πρέπει να αναμένουμε λοιπόν ισχυρές επικρίσεις ε, επί του θέμα κατά τη της του Δεκεμβρίου. Ευχαριστούμε. Τέλος ο κύριος Κελόμου. Σας με ενέπνευσε κύριε Υπουργέ η ρεαλιστική και ολοκληρωμένη προσέγγιση σας στην Ευρωπαϊκή Αμυντική Πολιτική και η προειδοποίησή σας για τα θέματα τα οποία είναι κοινά σε όλους μας. Είμαι απογοητευμένος επειδή δεν έχουμε δράση από κοινού και επίσης ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός ε, έχει μειωθεί, έχει περικοπεί. Στο Βίλνιους εκφράσατε τις ελπίδες σας ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Δεκέμβριο θα υπάρξει μια νέα δέσμευση για το δυναμικό, το ευρωπαϊκό και ε, ήθελα να σας ρωτήσω εάν αυτό θα εγκριθεί από το ε, ε, Συμβούλιο Υπουργών αν αυτό πραγματικά μπορεί να γίνει. Έχετε δεσμευτεί έντονα ε, στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού δυναμικού. Αλλά μέχρι τώρα θα έλεγα ότι τα φαινόμενα, η πραγματικότητα δείχνει ότι δεν υπήρξε πραγματική δέσμευση. Εσείς ξέρετε σαφώς τι σημαίνει μια πολιτική, ένας πολιτικός καλοπισμός, μια βελτίωση. Εγώ πιστεύω πολιτικά Μπορούμε να βελτιώσουμε την εικόνα και δεδομένου ότι γίνονται πάρα πολλές ε, επιχειρήσεις στο διάστημα, στο μέσο των ευρωπαϊκών ενεργειών, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τις ε, μειονοτικές ομάδες των ρωσικών πολιτών στην επικράτειά μας. Ο κύριος Γιάννης, θέλετε να κάνετε μια ερώτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είχα ζητήσει αρχικά το λόγο, γιατί συνήθως όταν συμφωνώ με τον ομιλητή, ε, για εξοικονόμηση χρόνου, να βοηθήσω και τον Υπουργό να προλάβει το τρένο του. Γι' αυτό δεν σκόπευα να πάρω το λόγο. Συμφωνώ λοιπόν με αυτά που είπε. Όμως τελικά ζήτησα το λόγο γιατί κατάλαβα ότι η μόνη φωνή που θα ακουστεί από τον Νότο θα είναι δικιά μου. Εντάξει, μπορούμε να πούμε βέβαια ότι η Γαλλία είναι και νότος και κέντρο και βορράς, αλλά εν πάση περιπτώσει από την Νότια Ευρώπη ήθελα να έχει ακουστεί και μια τέτοια φωνή. Εσείς είσαστε από μια χώρα του βορρά, εγώ είμαι από μια χώρα του νότου. Η πολιτική, η κοινή ασφάλεια και άμυνας είναι καλό να γίνεται σε συνεργασία του βορρά και του νότου. Οπότε μόνο να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ και να πω ότι συμφωνώ με όσο είπαν οι προλαλήσαντες και ιδιαίτερο ο Πρόεδρος Δαντζάν για την Λευκή Βίβλο κυρίως. Ευχαριστώ. Ο Υπουργός. Ευχαριστώ συνάδελφοι για όλες τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις που έχω μέχρι τώρα. Κύριε Γκέλλερ, όσον αφορά τις μάχημες ομάδες και τη νέα προσέγγιση, πιστεύω ότι πρέπει να ορίσουμε σαφέστατα τις φιλοδοξίες μας, τις επιδιώξεις μας και να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ομάδες δεδομένου ότι υπήρχε έντονος ε, αντίκτυπος ε, και αποτελέσματα από παρόμοιες ομάδες, μάχημες δηλαδή, άλλων χωρών. Πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε με την καλύτερη δυνατότητα και Βεβαίως ε, η εδραίωση της ειρήνης στην Ευρώπη είναι η μεγαλύτερη μας επιτυχία. Όμως πρέπει να βρούμε τρόπους να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις μάχημες ομάδες. Αύριο έχουμε ένα σεμινάριο με τους εταίρους μας, με τους της ομάδας μας για τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τις ε, ομάχημες εργασίες, ε, τις ομάχημες ομάδες με συν συν ή πλην ε, διότι αυτές εμπίπτουν στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι θα δώσουμε ένα σωστό μήνυμα για το μέλλον εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, αποφασίσει μία αναθεώρηση του δυναμικού αυτού εν ώψη νέων απειλών και νέων δυνατοτήτων που προσφέρονται, που παρουσιάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τη χρηματοδότηση τώρα, η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ της χρηματοδότησης από τα κράτη-μέλη και της χρηματοδότησης από πλευράς Ένωσης. Αυτό θα μας δώσει μια πραγματικά ισόρροπη κατάσταση και θα μπορέσουμε να πούμε ότι και τα κράτη-μέλη συνδράμουν και η Ένωση αυτή καθεαυτή βοηθά επίσης. Πολλοί ανέφεραν και το πρόβλημα της μεταφοράς, των μεταφορών. Ε, αυτό συμπίπτει και με <laughs> την ε, στάση μας ή τη στάση του μεγάλου γείτονα έναντι ημών. Ε, θα ήθελα να γίνουν και αυτοί να, μέλη ή να τέλος πάντων ε, κατανοήσουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συμμετάσχουν σε κοινέ ε, επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ. Ε, αλλά θα πρέπει να συνεργαστούμε και τις άλλες γειτονικέ χώρες, τις ε, από την Ουκρανία, τη Γεωργία, ε, ε, εκτός των Αμερικανών φίλων δηλαδή. Έγινε μία προσπάθεια συγκερασμού της, των ευρωπαϊκών αποστολών. Και όσον αφορά τη συνάντηση στο Βίλνιος το Νοέμβριο, η γυτνίαση με ανατολικές χώρες και η ανατολική πολιτική γειτονίας καλύπτει ε, και την αποδοτικότητα της πολιτικής διασφάλισης ενέργειας, ενεργειακών αναγκών, μαζί με την ασφάλεια. Όπως σας είπα, οι στρατιωτικές δυνάμεις, το στρατιωτικό σκέλος είναι το σκέλος που καταναλώνει την περισσότερη ενέργεια. Και αυτό βεβαίως έχει ένα αντίκτυπο στο κλίμα. Ε, αν δείτε τα θέματα αυτά, τα μελετήσετε πιο πολύ σε βάθος, θα διαπιστώσετε ότι προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους πόρους πιο αποτελεσματικά, λαμβάνοντας υπόψη και την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον. Τώρα το θέμα του κυρίου Saugumo ε, ir του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, όσον αφορά ε, την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, έχουμε πολύ καλή εμπειρία μέχρι τώρα η συνεργασίας με τις στρατιωτικές υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου. Ειδικά Α, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ε, μάχημες ομάδες στην Ευρώπη. Ε? Όσοι ε, γνωρίζουμε τα δεδομένα των ομάδων αυτών, των οποίων που επικεφαλής είναι ε, στρατιωτική του Ηνωμένου Βασιλείου, θα έλεγα ότι λειτουργούν πάρα πολύ καλά ένα θαυμάσιο παράδειγμα εφόσον μπορέσουμε να εδρώσουμε μία καλύτερη συνεργασία για τις κοινέ επιχειρήσεις θα πρέπει οπωσδήποτε να αποτανθούμε και στις Ηνωμένε Πολιτείε και να συνεργαστούμε και με εκείνους. Παραδείγματο χάρη, Ηνωμένε Πολιτείε επί δεκαετίες μας έδειξαν, μας δίνουν το παράδειγμα εδώ και δεκαετίες για το πώς λειτουργούν και χρηματοδοτούν τις δικές τους στρατιωτικές αποστολές. Πιστεύω ότι έχει φτάσει ο χρόνος για την Ευρωπαϊκή Ένωση να καλύψουμε ήδη με τις δικές μας δυνάμεις την ασφάλεια και την άμενα σε πολύ μεγαλύτερο εύρος από ό,τι στο παρελθόν. Ε, δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε με το τεράστιο στρατιωτικό δυναμικό θα είναι οι μόνε που θα μας προστατεύσουν. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και την υποστήριξή σας κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Πιστεύω ότι η πλαστική χειρουργική θα με βοηθήσει όχι μόνο στην βελτίωση της εμφάνισης αλλά και στην, στη βοήθεια προς μικρά, ιδίως σε μικρά παιδιά και βρέφη για να όχι μόνο να είναι πιο όμορφα αλλά να είναι και η ζωή τους πιο ευχάριστη, πιο καλή ποιοτικά. Πιστεύω ότι το Συμβούλιο Κορυφής όταν μιλάμε για τις φιλοδοξίες τις δικές μας, της Ένωσης, και επειδή είναι δύσκολο να προβλέψουμε το μέλλον, πιστεύω ότι το, Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα μας καλύψει, θα μας υποστηρίξει. Όσον αφορά τις, τις ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, πιστεύω ότι η Ρωσία, όπως κάθε άλλη χώρα, έχει το δικαίωμα να ενεργήσει όπως θεωρεί σωστό. Αλλά οι ενέργειές της πρέπει να είναι διαφανείς, και ε, μη απειλητικές ε, προς γειτονικέ χώρες. Εδώ εμείς έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση ε, από ό,τι έχει η Ρωσία σε αυτά τα θέματα. Κατανοούμε τις αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις, ότι αποτελούν ένα μικρό μέρος όλης της άσκησης και δεν νομίζουμε, δεν πιστεύουμε ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα είναι βαριά στρατιωτικής φύσης. Ο, τώρα, ο, θα ήθελα να συνεχίσουμε την ε, συνύπαρξή μας με φιλικό και ειρηνικό τρόπο με τη Ρωσία. Αλλά ε, εμείς θέλουμε να έχουμε φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία. Εγώ γεννήθηκα εκεί, δεν θα έλεγα την, ε, το, το, πάτριο έδαφος, η, η πατρική μου χώρα, αλλά θα πρέπει η χείρα φιλίας που τίνουμε εμείς προς τη Ρωσία να βρίσκει ανταπόκριση και από την άλλη πλευρά. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Τηρήσαμε το χρόνο μας, τον λίγο που είχαμε στη διάθεσή μας, μια χαρά. Παρ' όλα αυτά, συζητήσαμε επί της ουσίας και σε βάθος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα δούμε τι θα βγει από τις διασκέψεις κορυφής. Γιατί αναφερθήκαμε και στη διάσκεψη για την ε, ανατολική εταιρική σχέση. Η διάσκεψη πάντως για την άμυνα είναι κάτι αρκετά σπάνιο και γι' αυτό και περιμένουμε πολλά. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς εδώ. Να μην έχουμε προσδοκίες που να είναι ψευδέστηση, όχι, να είμαστε ρεαλιστές για να έχουμε κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτό χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε να προδεύουμε στην κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Καλό σας ταξίδι στο Λονδίνο. Υπενθυμίστε στους ομολόγους σας Βρετανούς ότι πολύ θέλουμε να τους έχουμε κάποια μέρα εδώ. Είμαστε πολύ περίεργοι και πολύ μας ενδιαφέρει η θέση που θα πάρει τελικά το Λονδίνο στη διάσκεψη αυτή. Γιατί εμεί εδώ βλέπετε είμαστε πολλοί που πιστεύω ότι μια πραγματική πολιτική άμυνας δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς μία από τις κύριες δυνάμεις στον τομέα της άμυνας στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Στο Πανεδίνο. Euh, Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Θα ακολουθήσει μια ανταλλαγή απόψεων για μια αποστολή της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελάχιστα γνωστής, αλλά πολύ σημαντικής και η οποία αφορά τη Λιβύη. Σας παρακαλώ λοιπόν αρχικά να Μα συγχωρέσετε για την απουσία του αρχηγού της αποστολής, του συνταγματάρχη Αρτικάινεν, ο οποίος χρειάστηκε να παραμείνει στη Λιβύη λόγω των γεγονότων της πέρασμενης εβδομάδας. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σταθής. Γι' αυτό θεωρήθηκε προτιμότερο να βρίσκεται ο αρχηγός αποστολής ε, στη Λιβύη. Για την ανταλλαγή απόψεων έχουμε μαζί μας τον κύριο Hans Jörg Haber, διοικητή στρατιωτικών επιχειρήσεων και διευθυντή τη EPCC με τον κύριο Χάμπερ θα σας ενημερώσουμε για την κατάσταση στην Τρίπολη δεδομένης της αβεβαιότητας την οποία σας ανέφερα αλλά και πιο συγκεκριμένα για αυτή την αποστολή συνδρομής για τη φύλαξη των συνόρων, την UBAM. Ε, όπως γνωρίζετε αυτή η εντολή για τη Λιβύη ανατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν καν τελειώσουν οι σειράξει, διότι στη διάσκεψη του 2011 ήδη στη διάσκεψη του Παρισιού υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών έγινε κάποια κατανομή καθηκόντων όσον αφορούν τα ζητήματα ασφάλειας της Λιβύης και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αναφέρει ότι μπορούσε να εργαστεί για το θέμα της συνοριοφυλακής. Πολλές δυσκολίες συναντήσαμε έκτοτε. Η πρώτη και κυριότερη ήταν η απουσία καθαρά καθορισμένων συνομιλητών στην ίδια τη Λιβύη ώστε να μας εκφράσουν τις απόψεις του κράτους και για να επισημοποιηθεί η μορφή της συνεργασίας αυτής. Ε, συνεχίζουν να υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες από όσο έχω καταλάβει. Υπάρχει κάποια θεσμική αστάθεια που καθιστά ιδιαίτερα ευαίσθητη τη διατύπωση των αναγκών από τις λιβικές αρχές. Συχνά αληθεύει το Κοινοβούλιο, επικρίνει τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση αυτής της αποστολής, αλλά θα έχει ενδιαφέρον να μας αναφέρετε εσείς ε, τα συγκεκριμένα σημεία παρουσίας σαν προβλήματα. Ξεκίνησε η αποστολή τον Μάιο του 2013, αν δεν κάνω λάθος, κάποιος αριθμός ε, προσωπικού αναπτύχθηκε στη Λιβύη αλλά σε περιορισμένο αριθμό. Γι' αυτά θα θέλαμε να μας ενημερώσετε. Πρόκειται για μια αποστολή σχετικά άγνωστη η οποία χρήζει διευκρίνηση. Και κυρίως πρέπει να δούμε ποιες είναι οι προοπτικές. Κατά πόσο μπορούμε εύλογα να ελπίζουμε ότι αυτή η αποστολή θα καταλήξει κάτι συγκεκριμένο σε εποχές ε, όπου οι ανάγκες ε, είναι ιδιαίτερα επιτακτικές και λόγω των γεγονότων που βλέπουμε στη Λιβύη αλλά και για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό των μεταναστευτικών ροών που πάλι βρίσκονται στο προσκήνιο της επικαιρότητα. Και όπως παρατηρήσαμε το πρόβλημα ξεκινάει ήδη από τα νότια σύνορα της Λιβύης πριν φτάσει στη Μεσόγειο. Υπάρχει λοιπόν και το θέμα αυτό των νότιων σύνορων με το οποίο πρέπει να ασχοληθεί η αποστολή Ιουμπάμ. Κύριε Εύερ, σας δίνω το λόγο και θα συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι, να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρου του αρχηγού αποστολή του κ. Χαρτικάινεν που δεν βρίσκεται εδώ. Όπως γνωρίζετε, Υπήρξε η απαγωγή του Πρωθυπουργού την περασμένη Πέμπτη και η ελευθέρωση του που επακολούθησε και το γεγονό έλαβε χώρα στο ίδιο το ξενοδοχείο που βρίσκεται και η αποστολή. Συνεπώ, ε, παρέμεινε ο αρχηγό αποστολή ε, επί τόπου για να εξετάσει από κοντά τα συμπεράσματα που μπορούμε να εξάγουμε από το γεγονό αυτό. Σα ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την δυνατότητα να σα μιλήσω για την αποστολή και όπως είπε ο κύριος Πρόεδρος είναι μια ελάχιστα γνωστή αποστολή που όμως ε, θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη προσοχή και μόνο λόγω των προσδοκιών που υπάρχουν με τα, από τα θλιβερά γεγονότα που έλαβαν χώρα στη Μεσόγειο. Και θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να σας αναφέρω κάπως τις προσδοκίες, ε, τις δυνατότητες που διαβλέπουμε εμείς ε, μακροπρόθεσμα. Όσον αφορά την απαγωγή του Πρωθυπουργού, συμπεραίνουμε αστάθεια της πολιτικής κατάστασης στη Λιβύη. Η μεταβατική διαδικασία χρειάζεται χρόνο. Το έργο της κυβέρνησης παρεμποδίζεται από τις πρόσφατες απεργίες του σημεία παραγωγής πετρελαίου και ο αργός ρυθμός πρόθεσης των συνταγματικών μεταρρυθμίσεων δημιουργεί ενοχλήσεις και η έλλειψη ελέγχου σε θέματα ασφαλείας ε, δυσκολεύει τον πολιτικό ρόλο των ε, όσων ασχολούνται με την ασφαλεία στη Λιβύη. Η πρόσφατη απαγωγή του Πρωθυπουργού έγινε από την ε, ομάδα των Σαλαφιστών που υποστηρίζονται από την ε, μουσουλμανική αδελφότητα και επικρίθηκε σημαντικά ε, στο Κοινοβούλιο της Λιβύης. Μετά από την απελευθέρωσή του, ο Πρωθυπουργό δήλωσε ότι οι πολιτικοί του αντίπαλοι προσπάθησαν να προβούν σε αυτή την ενέργεια για να τον αναγκάσουν να παραιτηθεί εξαναγκάζοντας ψήφο εμπιστοσύνης στο Εθνικό Κογκρέσο. Η πολιτική λοιπόν και η ασφάλεια είναι αλληλένδετες στη σημερινή Λιβύη. Σε μεγάλο βαθμό. Η κατάσταση της ασφάλειας ειδικότερα υποβαθμίζεται και οι βιοπραγίες αυξάνονται. Μετά από την ανάπτυξη της αποστολής το Μάιο του 2013, αναμφίβολα η ασφάλεια έχει υποβαθμιστεί. Αυτό σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την εσωτερική πολιτική και είδαμε πολιτικές δολοφονίες στρατιωτικών αστυνομικών. Η διεθνή κοινότητα επίσης ε, αποτέλεσε πρόσφατα στόχο παρότι όχι σε μεγέθη συγκρίσιμα όπως αυτά που βλέπουμε στο Αφγανιστάν. Η δυσαρέσκεια με την κυβέρνηση και το Εθνικό Κογκρέσο και την εθνική ασφάλεια και η αργή διαδικασία μετάβασης, όλα αυτά μπορεί να επηρεάσουν και τη διεθνή παρουσία. Ο Λίβες Πρωθυπουργό και η κυβέρνηση στο σύνολό τη συνέχισαν να ζητούν την αρρωγή της διεθνούς κοινότητας για τη σταθεροποίηση της χώρας και για την ανάπτυξη της ασφάλειας στη Λιβύη. Μεταξύ άλλων, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη τόνισαν τη συνεχή του υποστήριξη για την κυβέρνηση της Λιβύης, ενώ καλούν όλα τα μέρη, τα διαφρόμενα τη Λιβύης να βοηθήσουν στην οικοδόμηση μιας ισχυρή και σταθερής ε, χώρας. Ειδικότερο όσον αφορά την ασφάλεια τη αποστολής. Η γενική κατάσταση της ασφάλειας στη Λιβύη έχει ληφθεί υπόψη στην κατάρτιση μέτρων μετριασμού που έλαβε η αποστολή και που υλοποιούνται σήμερα. Ειδικότερα, ο ρυθμός ανάπτυξης του σημερινού προσωπικού έχει προσαρμοστεί. Αυτό σημαίνει καθυστερήσει σύμφωνα με την εξελισσόμενη κατάσταση στη χώρα. Τα μέλη της Επιτροπής ε, μπορεί να γνωρίζουν τις λεπτομέρειες του, της απαγωγής του Πρωθυπουργού. Αυτό έγινε στο ίδιο ξενοδοχείο με εκείνο που διαμένει η αποστολή. Το ξενοδοχείο Κορίνθια παρόλα αυτά θεωρείται η πιο ασφαλής τοποθεσία για την αποστολή στην Τρίπολη. Το συμβάν αυτό υπογραμμίζει πόσο επίγοντα είναι τα μέτρα που πρέπει να λυθούν ώστε να μεταφερθεί σε ένα μόνιμο κέντρο η αποστολή. Αλλά φυσικά οι προμήθειες παρεμποδίζουν την οριστικοποίηση των εργασιών και καθυστερούν τη μεταφορά της αποστολής. Παρακολουθούμε την κατάσταση σε συντονισμό με την Εταιρεία Παροχής Ασφάλειας, με την Αντιπροσωπεία, με τις πρεσβείες των κρατών μελών και άλλους διεθνείς παραγόντε που είναι παρόντες εκεί, όπως ειδικότερα τα Ηνωμένα Έθνη. Οι διευθετήσεις ασφαλείας επανεξετάζονται διαρκώς, αλλά το περιθώριο προσαρμογής τους, δεδομένων των σημερινών περιστάσεων και των διαδικασιών που υπάρχουν, είναι περιορισμένο όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Εκεί τα πράγματα είναι κάπως πιο αισιόδοξα. Παρά την ασταθή πολιτική και την αστάθεια της ασφάλειας και την γενικότερη αβεβαιότητα και παρά τη φάση οικοδόμησης την οποία βρίσκεται η αποστολή έχουν ληφθεί αποφασιστικά βήματα για την υλοποίηση της εντολής. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 45 μέλη του διεθνούς προσωπικού ενώ έχει επιτραπεί ε, η επάνδρωση με 111 μέλη. Συνεπώς λιγότερα από τα μισά. Η αποστολή υποστηρίζει την ανάπτυξη της ομάδας εργασίας διαχείρισης των συνόρων που δραστηριοποιείται υπό το γραφείο του Πρωθυπουργού και που συντονίζει τη συνεργασία των οργανισμών διαχείρισης των συνόρων της Λιβύης. Η αποστολή είναι παροχή συμβουλών και η συνεργασία σε αυτή την ομάδα για τη βελτίωση της στρατηγικής ε, διαφύλαξης των συνόρων. Παρότι το γραφείο του Πρωθυπουργού και η ομάδα εργασία για τη φύλαξη των συνόρων είναι οι κύριοι συνομιλητέ για την αποστολή, έχουμε καταφέρει να διευρύνουμε το δίκτυο αυτό και να έρθουμε σε επαφή με ομολόγου εντό των θεσμικών οργάνων τη Λιβύης ώστε να μετριάσουμε την αβεβαιότητα τη πολιτική κατάσταση με τακτικέ ανταλλαγέ ε, απόψεων με διάφορου συνομιλητέ. Το γεγονός ότι η αποστολή παρέχει συμβουλές ε, για την ε, ανοικοδόμηση ενός οργανισμού όπως του Λιβικού Οργανισμού Διάσωσης μαρτυρεί τη σημαντική διάσταση που έχει λάβει η αποστολή μας εκεί καθώς και την εμπιστοσύνη των τοπικών αρχών επίσης ε, δείχνει τα επιτεύγματα και τις προκλήσεις που απομένουν ενώπιον μας η αποστολή υποστηρίζει τους Λίβιους στις προσπάθειές τους για αύξηση των τεχνικών δεξιοτήτων των ατόμων που εργάζονται στις υπηρεσίες φύλαξη των συνόρων μέσω ενός προγράμματος κατάρτισης και καθοδήγησης. Αυτό εν το χρόνο θα ενισχύσει την ικανότητα των λιβικών αρχών να χειριστούν τα συνοριακά εγκλήματα όπως την μεταφορά, την παράνομη μεταφορά, το εμπόριο ανθρώπων και την παράνομη μετανάστευση. αλλά απομένουν και άλλες εξελίξεις, χρειάζεται και περισσότερη στελέχωση των αποστολών, καθώ και μαζί με την κατάρτιση. Η αποστολή βρίσκεται στην Τρίπολη, αλλά βρίσκεται εκεί για να βοηθήσει τη φλεξόνα των σύνορων της Λιβύης. Έχει διεξάγει ε, επισκέψεις μελέτη στα σύνορα με την Τουνησία, στον Καραμές, στο σύνορα μεταξύ Λιβύης, Τουνησίας και Αλγερία, στο νοτιότερο μέρο της Τινησίας, στο σύνολο της Μισράτα, καθώς και στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μιστάβα στην νότια πλευρά που ήταν σημαντικό στην κρίση στη Λιβύη. Οι δικαιούχοι αυτής της βοήθειας είναι οι συνοριοφύλακες, η συνορική αστυνομία, η ενάρια ασφάλεια και η ασφάλεια των αεροδρομίων και των λιμένων. Εμείς εκτιμάμε ότι είναι εφικτή η αποστολή της Γιουμπάμ, αλλά το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Και δυστυχώ δεν ελέγχουμε εμεί αυτό το χρονοδιάγραμμα. Θα εξαρτηθεί από την συνεχώ μεταβαλλόμενη κατάσταση τη ασφάλιση. Οι περιορισμένε δυνατότητε απορρόφηση στη Λιβύη επίση προκαλούν καθυστερήσει στην υλοποίηση τη εντολή τη αποστολή. Αυτά ήθελα να σα πω. Ευχαριστώ για την προσοχή σα και είμαι στη διάθεσή σα να προσπαθήσω να απαντήσω τις ερωτήσεις σας, αν έχετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ερώτηση, σχόλιο, αλλά σκέφτηκα αυτό που είπατε για την ε, τοποθεσία, για το μέρος. Πρώτα απ' όλα σημειώνω ότι ο Πρωθυπουργό Λίβιο όπω και η αποστολή της Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο ξενοδοχείο Κορίντια, έτσι. Κάτι λέει αυτό. Ένας πρωθυπουργός που ζει στο ξενοδοχείο, ναι, αλλά τι γίνεται με την ασφάλεια στην πόλη. Έχουμε τη συνήθεια, δυστυχώς θα έλεγα, να διαπιστώνουμε ότι οι μη στρατιωτικές μας αποστολές που αναπτύσσονται σε δύσκολες περιοχές δεν έχουν πάντα στη διάθεσή τους την κατάλληλη υποδομή διαχείρισης η διαχείριση, για λόγους που εν μέρει αναφέρατε, που είναι διοικητικοί, που έχουν να κάνουν με προσφορές που γίνονται από την ίδια τη χώρα, οι αποστολές δεν διαθέτουν ούτε τα κτίρια, ούτε τα οχήματα, ούτε τα μέσα επικοινωνία στα κατάλληλα. Μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση α, τα βγάζει πέρα, λίγο αυτοσχεδιάζοντας, ελπίζοντας ότι μετά από μερικούς μήνες η κατάσταση θα διορθωθεί. Όμως, έτσι επικίνδυνη που είναι η κατάσταση στη Λιβύη σήμερα, αναρωτιέμαι. Είναι επιθυμητό, είναι λογικό, σωστό να αναπτύσσεται προσωπικό σε ένα ξενοδοχείο χωρίς να έχουμε ακόμα τους κατάλληλους χώρους για να υποδεχτεί μία αποστολή και να παρέχει έχει ασφάλεια. Ε? Έπειτα υπάρχουν και μεταφορές, επικοινωνίες που χρειάζονται καλύτερη, ε, να είναι πιο, σε πιο καλή κατάσταση από αυτά που έχουμε σήμερα στη Λιβύη. Η ασφάλεια του προσωπικού λοιπόν, γιατί ακόμα και για στρατιωτικές αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σκέφτομαι εκείνη στο Μαλί, την εκπαιδευτική στο Μαλί. Και εκεί η συζήτηση ήταν τεράστια για την προστασία των δυνάμεων. Δηλαδή και στρατιωτικοί οι οποίοι πάνε σε μια περιοχή που δεν είναι πια σε εμπόλεμη κατάσταση, έτσι. Γιατί δεν ήταν εκεί που γίνονταν οι μάχες. Παρόλα αυτά η Force Protection είναι ένα στοιχείο πολύ σημαντικό και σε εκείνη την περίπτωση. Εδώ λοιπόν ποιος διασφαλίζει την ασφάλεια των Ευρωπαίων μας που συμμετέχουν στην αποστολή αυτή. Γιατί δεν φαντάζομαι ότι είναι οι ίδιοι Λίβοι, οι στρατιωτικοί. Τι σιγουριά υπάρχει. Ερωτήσεις είναι αυτές που περνάνε από το κεφάλι μου. Και επί τόσο αφορά τις προοπτικές, γιατί εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι έχουμε ομάδα εργασίας για τη διαχείριση συνόρων, Αυτά που ακούμε, πληροφορίες που μας έρχονται όμως είναι ότι η ασφάλεια με πολλά εισαγωγικά, έτσι, των νοτίων συνόρων της Λιβύης ιδιαίτερα, στην Μισράτα κλπ, τα έχουν κάτι, κάτι μπα, κάτι επαναστατικές μονάδες, οι οποίες δεν θέλουν να είναι υπό τις διαταγές των, του τακτικού στρατού, τον οποίο δεν αναγνωρίζουν στο κάτω-κάτω. Οπότε εμείς με ποιους συνεργαζόμαστε. Με ε, στρατιωτικούς επίσημους που είναι στην Τρίπολη αλλά που δεν τους βλέπουμε απαραίτητα αλλού ή με ό,τι ε, δυνάμεις, μονάδες βρούμε επιτόπου. Με ποιους συνεργαζόμαστε. Όλα αυτά μου φαίνονται πολύ αόριστα και ασαφή. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Μίκαελ Γκάλερ τώρα. Ευχαριστώ. Και εγώ συμφωνώ με τον προλαλήσαντα. Οι ερωτήσεις αυτές <clears throat> βασίζονται στις προηγούμενες εξέσεις και αναφορές που είχαμε και όλες λένε, λένε ότι η κατάσταση χειροτερεύει και τελικά η Λιβύη τίνει να γίνει ένα ε, τελείως κατεστραμμένο και διαλυμένο κράτος. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω εάν αυτή είναι η κατάσταση και εάν αυτή η βάση εκκίνησης είναι πάρα πολύ μικρή για να μπορέσουμε να ενεργήσουμε. Μήπως θα πρέπει να διευρυνθεί καταρχάς στατιωτικά ε, αστυνομικά έτσι ώστε να μπορέσουμε να διευρύνουμε το δυναμικό ασφαλείας και να συμμετάσχουμε σε πολύ περισσότερο βαθμό στη διοργάνωση. Ε, κάποια έσοδα από τα, το πετρέλαιο το, τα παίρνει το κράτος. Υπάρχουν κάποια έσοδα, κάποιοι πόροι, αν και είναι περιορισμένοι. Αλλά το, θέμα είναι ότι η αστυνομία και ο στρατός ζητούν να, καταταγεί, ζητούν ε, να καταταγούν και συνεχεία όποιος κατατάσσεται φέρνει και το δικό του όπλο. Αναρωτιέμαι λοιπόν μήπως η, η βάση διαβούλευσης και δραστηριοποίησης πρέπει να είναι πολύ ευρύτερη από αυτή την στενή επιχειρησιακή βάση που έχουμε τώρα και αναφέρθηκαν ήδη γραφειοκρατικά εμπόδια όσον αφορά δημόσιους διαγωνισμούς κλπ. Αλλά αυτό αυτές οι μη στρατιωτικέ αποστολές ε, τα κράτη-μέλη τις θεωρούν εξαιρετικά ε, λαμπρή ιδέα, αλλά δεν εγκρίνουν την αποστολή προσωπικού. Ωραία όλα και καλά, αλλά χωρίς προσωπικό, είπατε 45 έχουν εγκριθεί από τον συνολικό αριθμό των 111. 45 είναι εκεί, ενώ θα μπορούσαν να είναι, έχουν εγκριθεί 111 θέσεις. Άρα λοιπόν τι μπορεί να γίνει με την άρνηση αποστολής προσωπικού. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν άλλε παρεμβάσει αυτή τη στιγμή. Κύριε Μάικλ Γκαρέλερ, μιλώντα για τη δέσμευση των κράτων μελών, ε, θυμάμαι μια άλλη ερώτηση. Τι γίνεται με τι διμερείς δεσμεύσει, διότι εδώ μιλάμε για τη συλλογική αποστολή τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο τη κοινή Πολιτική ασφάλειας και άμυνας, αλλά νομίζω ότι ορισμένα κράτη-μέλη, όπως νομίζω η Γαλλία, η Ιταλία, οι Βρετανοί, αναπτύσσουν τις δικές τους επαφές και τις δικές τους ε, πολιτικές όσον αφορά τα ζητήματα ασφαλής και τις σχετικές συζητήσεις με τη Λιβύη. Έχετε κάποια ενημέρωση, υπάρχει κάποιο είδους ε, έστω και ελάχιστο συντονισμός, ε, έστω και ενημερωτικός όσον αφορά τις ενέργειες των κρατών μελών που καμιά φορά μπορεί να έρχονται σε αντίθεση με τη συλλογική προσπάθεια της EUBAM. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όλα αυτά είναι πραγματικά πολύ ε, βάσιμες παρατηρήσεις. Ήμασταν πολύ υπερήφανοι ε, στην, για την αποστολή αυτή, όπως στην περίπτωση της ε, ε, ταχείας, ε, δύναμης ταχείας ανάπτυξης, η οποία όπου είχαν πετύχει, είχαμε θετικά αποτελέσματα, όπως στην περίπτωση του Νίγηρα. Το θέμα είναι ότι αυτή η αποστολή τώρα στο έδαφος μπορεί να προμηθευτεί ορισμένα πράγματα, έχουν εγκριθεί ορισμένες προμήθειες, αλλά όχι πέραν αυτών που ενέκρινε το τελευταίο συμβούλιο. Έχουμε τώρα ένα πολλά προσκόμματα. Εάν μπορούσαμε εξ αρχής να είχαμε τη δική μας βάση, το δικό μας συγκρότημα όπου θα στεγαζόταν η αποστολή, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερες επιτυχίες. Όμως υπάρχουν τρομερές καθυστερήσεις ε, στον προγραμματισμό και στην κατασκευή. Αυτό το καταλαβαίνετε. Είναι ευνόητο. Το ίδιο ισχύει και στον τομέα της ασφάλειας. Ε, πρέπει να ξαναγίνει προκήρυξη της σύμβασης ε, αυτό γίνεται συχνά σε όλο το πλαίσιο διαδικασίας δημοσίων συμβάσεων. Έπρεπε να ξαναγίνει ο διαγωνισμός, να ξαναγίνει η σύμβαση, να υπογραφεί κλπ. κλπ. Όλα αυτά καθυστέρησαν ε, την διαδικασία, ε, διότι έπρεπε να γίνουν σεβαστές οι νέες διαδικασίες. Εμείς τα πρώτα προτιμούσαμε βεβαίως να είχαμε κάτι καλύτερο και νωρίτερα το θέμα λοιπόν παραμένει κρεμές. Και εμείς στις αποστολές της κοινή πολιτικής άμυνας και ασφάλειας ε, πρέπει να ε, έχουμε τη δυνατότητα να διενεργούμε αυτές τις, ε, τους μειοδοτικούς διαγωνισμούς και τις αναθέσεις πολύ ταχύτερα και πολύ πιο αποτελεσματικά, να είμαστε πολύ πιο ευέλικτοι και πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι εδώ δεν ε, εργαζόμαστε σε μια ε, τέλεια αγορά όπως την εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά σε μια σταθή ε, επικίνδυνη αγορά όπως τη Λιβύη. Εάν και, και πάρα πολύ ενδιαφερόμενοι να αναλάβουν τις συμβάσεις, τα έργα αυτά ε, παρετούνται όταν δουν τις συνθήκες που επικρατούν στο έδαφος και τις προδιαγραφές. Ε, όσον αφορά τώρα το θέμα της ε, προστασίας των δυνάμεων προστασίας είχαμε τα, ίδιο, τα ίδια προβλήματα όπως το Αφγανιστάν. Τα κράτη-μέλη είπαν ότι δεν θέλουν ε, τις ε, στρατιωτικές ή αστυνομικές τους δυνάμεις να προστατεύουν κάθε μέλος της αποστολής για βάση της εντολής, ε, δυνάμεις προστασίας δηλαδή. Άρα πρέπει να βασιστούμε σε ιδιωτικές υπηρεσίες παροχής ασφάλειας ε, ε, που πρέπει να τηρούν τον ε, κώδικα συμπεριφοράς της Λοζάνης. Γενικά έχουμε καλή εμπειρία από τις εταιρείε παροχής ασφάλειας. Όχι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και περισσότερα πράγματα. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε και άλλες εταιρείε για υπηρεσίες ασφάλειας, παραδείγματο χάρη στο Αφγανιστάν, όπου υπάρχουν πάρα πολλέ εσωτερικέ επιθέσει, δηλαδή από τις ε, δικές μας ε, δυνάμεις ε, σε στελέχη που υπηρετούν εκεί. Πρέπει λοιπόν και να προσφεύγουμε σε ιδιωτικές εταιρείες και πρέπει να βασιζόμαστε και στην ε, υποστήριξη από τις τοπικές δυνάμεις, οι οποίες βεβαίως δεν είναι πάντοτε φερέγγιες, όπως είδατε και στην περίπτωση της απαγωγής του Πρωθυπουργού. Επίσης μην ξεχνάτε ότι ε, υπάρχει και το ε, η φιλετική διάσταση. Όχι, δεν έχουμε υποστήριξη από όλες τις φυλές ε, υποτίθεται ότι ο έλεγχος εκεί επιβάλλεται μέσω της συνένεσης και της πολιτικής διαδικασίας. Ε, εμείς παρέχουμε συμβουλές για το τι μπορεί να κάνουν τώρα και τι μπορεί να κάνουν στο μέλλον για την εδραίωση του ελέγχου. Δεν έχουμε καμία εντολή ε, σχετική με αυτές τέτοιους παρεμβάσεις ούτε μπορούμε να στεκόμαστε εκεί στα σύνορα και να είμαστε παρόντες όταν εκτελούν την εργασία τους. Μόνο συμβουλευτικές δραστηριότητε μπορούμε να προσφέρουμε. Και τώρα όσον αφορά την, ε, το αν η Λιβύη είναι ένα κράτος πλήρους αποτυχίας ε, αυτή τη στιγμή το ανώτατο επίπεδο εξουσίας, τα ανώτατα στελέχη θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας με ενθουσιασμό. Αλλά αυτό δεν τους έχει εμποδίσει να ε, δεν, όλες αυτές οι δυσκολίες και τα προβλήματα δεν τους έχουν εμποδίσει να συνεργαστούν επιτυχώς με την αποστολή. Βεβαίως υπάρχουν πολλά προβλήματα πέραν της, των συνόρων και τη διαχείριση των συνόρων και της ε, παροχή συμβουλών και βοήθειας. Όμως δεν έχουμε και τις δυνατότητες να δράσουμε ε, περισσότερο. Έχουμε, είμαστε πάρα πολύ περιορισμένοι στα μέσα και στους πόρους που έχουμε και όσο περισσότερο εμφανές γίνεται το πολιτικό πρόβλημα τόσο περισσότερο αυξάνεται ο κίνδυνος επιθέσεων. Έχουμε ήδη όπως σας είπα το, το καυτό πρόβλημα των εσωτερικών ελέγχων δηλαδή να ελέγχουμε εσωτερικά τις υπηρεσίες μας και ε, αυτή αυτή στιγμή ε, πρέπει να επικεντρωθούμε στο στόχο μας που είναι η σωστή λειτουργία της αποστολής. Να αντιμετωπίσουμε την παρούσα κατάσταση ασφαλείας ως είναι, πρέπει να μεταφέρουμε τις εγκαταστάσεις μας σε μια μόνιμη βάση, μόνιμη εγκατάσταση και να ελπίζουμε σε μια καλύτερη κατάσταση ασφαλείας. Το ερώτημα τώρα του ελιπούς ε, προσωπικού ε, από πλευράς κρατών μελών δεν αφορά τη Λιβύη. δεν έχουμε ακόμα ζητήσει περισσότερο προσωπικό διότι δεν έχουμε και τη δυνατότητα από τη λιβικής πλευράς να προσλάβουμε διότι είναι αυτό που σας είπα το θέμα της ασφάλειας δεν μπορούμε να παράσχουμε την απαραίτητη ασφάλεια δεν είναι λοιπόν το ελληπές προσωπικό ε, θέμα των κρατών μελών ή έλλειψη από πλευράς κρατών μελών να παράσουν την εμπειρογνωμοσύνη. Ίσα ίσα τα τελευταία χρόνια είχαμε περισσότερες αιτήσει ε, περισσότερε προσφορέ από τα κράτη-μέλη. Ορισμένε φορέ δεν είναι μόνο η χρηματοδότηση, αλλά για την των στο Νότιο Σουδάν, παραδείγματο χάρη, μα λείπουν οι εμπειρογνώμενε Έχουμε προβλήματα με, με τον, τον εξοπλισμό, με τα εξοπλιστικά ε, ε, με τα συστήματα που χρησιμοποιούμε, τον εξοπλισμό, μηχανήματα κλπ. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Αλλά τα κράτη-μέλη γενικά διαθέτουν επαρκές προσωπικό. Επίσης, ορισμένες φορές ε, ε, ε, αποστολές όπου επικεφαλής είναι γαλλικά, στελέχη από τη Γαλλία, δεν υπάρχουν αρκετοί γαλλόφωνοι και παρεμφερεί προβλήματα. Αλλά υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, αρκά ικανοποιημένη με την γενική προθυμία των κρατών μελών να υποστηρίξουν υποψήφιους, ορισμός τους βεβαίως διαφέρει πολύ σημαντικά από κράτος σε κράτος και δεν λέω ότι το βάρος το φέρουν ισότιμα όλα τα κρατημέλη, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Νομίζω ότι απάντησα στις περισσότερες ερωτήσεις ε, όσον αφορά τις διμερείς πτυχές. Η αποστολή είναι ακόμα, βεβαίως έχει επαφές με την πρεσβεία. Νομίζω τρία μέλη, τρία στελέχη έχουν μείνει από τα δέκα που υπήρχαν. Γενικά πιστεύουμε ότι έχουμε μια σωστή ενημέρωση για το τι προγραμματίζουν από πλευράς πρεσβείας. Ωραία λοιπόν, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ωραίο βέβαια ομολογώ ότι βρισκόμαστε σε μια παράδοξη κατάσταση. Λυπάμαι που η Άννα που ήταν η συγγήτρια της ΑΦΕΤ για τη Λιβύα και που βρισκόταν στη Λιβύη πριν από δέκα μέρες, μόλις δεν είναι μαζί μας σήμερα. Έχουμε προσπαθήσει και πιέσει για να υλοποιηθεί επιτέλους κάτι διότι αναμφίβολα υπάρχει ανάγκη. Ταυτόχρονα έχουμε και κάποιους ενδιασμούς όσον αφορά αυτή την αποστολή η οποία σε μεγάλο βαθμό παραμένει αόριστη λόγω της επιτόπου κατάστασης. 45 στους 110 που έχουν προβλεφθεί δεν είναι πολύ μέλη του προσωπικού ε, αλλά θα ήθελα να δω και τι κάνουν κάθε μέρα όλοι αυτοί το να βρίσκονται στο ξενοδοχείο Κορίνθια και να εργάζονται με Λίβιους οι οποίοι τις μισές φορές δεν εμφανίζονται ή δεν δείχνουν ιδιαίτερη βούληση. Δεν μπορώ να φανταστώ τι ουσιαστικά αποτελέσματα μπορεί να έχει εργασία σε ένα τέτοιο περιβάλλον για να το σοβεί στο θέμα. Και εδώ ουσιαστικά σαν είναι πρόσχημα αποστολής αυτού, σαν να προσπαθούμε να πούμε ότι κάνουμε κάτι και η αλήθεια είναι ότι εμείς προσπαθούμε να ισχυριστούμε κάτι, ότι και εγώ τώρα αισθάνομαι άσχημα που επικρίνω κάτι τέτοιο, γιατί έχουμε επιμείνει ιδιαίτερα να γίνει κάτι στη Λιβύη, αλλά ε, έχω πολλά ερωτηματικά όσον αφορά την πραγματική υλοποίηση, την ουσία ουσιαστικά της αποστολής αυτής. Φυσικά κάποιοι λένε ότι είναι καλύτερα να βρισκόμαστε επί τόπου και αν ξεκινήσουν τα πράγματα να κινούνται θα ήταν πιο εύκολο να έχουμε ήδη άτομα επί τόπου αντί να ξαναξεκινάμε από τι Βρυξέλλε. Είναι βέβαιο αυτό, αλλά παρόλα αυτά εγώ διατρέω κάποιους ενδιασμούς σαν αφορά αυτή την αποστολή και την αποτελεσματικότητά της και το τι πραγματικά μπορεί να επιτύχει επί τόπου χωρίς επαναλαμβάνω να αμφιβάλλω καθόλου για τον επαγγελματισμό των υπευθύνων προγραμματισμού και όσων βρίσκονται εκεί, οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπίζουν εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις. Θα ήταν όμως ενδιαφέρον να ακούσουμε και από αυτούς κάποιες παρατηρήσεις για το τι έχει επιτευχθεί πραγματικά. Διότι 45 Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή στη Λιβύη ε, δεν είναι ανώδυνο ούτε πολιτικά ούτε οικονομικά για την Ευρώπη. Γι' αυτό έχω ενδιασμούς. Ενδιασμούς για την ουσία ουσιαστικά. Κυρία Νέτς. Ε, Πρόεδρε, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Χαμπέρ για τα όσα μας είπε. Δεν είμαι ειδική για τη Λιβύη, καθόλου δεν έχω πατήσει ποτέ το πόδι μου, οπότε δεν θα τολμούσα να πω πολλά επί του θέματος. Συμφωνώ βέβαια με τον πρόεδρο Ντανζόν για το εξή. Μέχρι τώρα είχαμε την τάση να υποτιμούμε τη δυσκολία και την πολυπλοκότητα των, της δουλειάς μας εκεί. Το κοσυφοπέδιο που είναι πολύ πιο περιορισμένο ε, από πλευρά τετραγωνικών χιλιόμετρων και η κατάσταση είναι και πιο απλή, αλλά αν δούμε τι προσπάθειες έγιναν και τι προσπάθειες πρέπει ακόμα να γίνουν για να διασφαλίσουμε μία βάση προκειμένου πιο αρμονικά και με περισσότερη σταθερότητα να εξελιχθεί η κατάσταση, φανταστείτε τι γίνεται με τη Λιβύη. Στη Βοσνία Ερζεγοβίνη επίσης, το ίδιο. Οπότε λέω ότι εδώ υποτιμήσαμε πάρα πολύ τις δυσκολίες για τη Λιβύη. Καταλαβαίνω τι λέτε, Πρόεδρε, αλλά τι θα έπρεπε να κάνουμε, να μην κάνουμε τίποτα, μήπως να περιμένουμε μέχρι να ξεμπερδευτεί λιγάκι το κουβάρι από μόνο του. Μερικές φορές γίνεται και αυτό. Ή μήπως, κάτι το οποίο όμως μου φαίνεται πολύ δύσκολο να το διανοηθεί κανείς, αν και μερικές φορές το έχουμε κάνει, μήπως θα έπρεπε να, να εγκαταστήσουμε κάτι σαν το πρόδρομο προξενικής αρχής, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Ειλικρινά, η δυσκολία της οικοδόμησης, της ανοικοδόμησης κρατικών δομών βασικών ε, στη Λιβύη, εκεί που δεν υπάρχουν, ε, που έπαψαν να λειτουργούν. Πώς θα το κάνουμε δεν θα έπρεπε να κρυβόμαστε απέναντι στις δυσκολίες, όχι, να τις αναγνωρίσουμε, γιατί κάθε φορά θα είναι περίπλοκη κατάσταση, κάθε φορά θα είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και κάθε φορά κακώς θα έχουμε ψευδεστήσεις και θα νομίζουμε ότι εμείς θα επαναφέρουμε τη δημοκρατία έτσι. Όχι, ούτε το κράτος δικαίου, ούτε τη δημοκρατία, ούτε τίποτα. Δεν είναι εύκολο. Ποια είναι η εναλλακτική. Είχαμε αποφασίσει κάποια στιγμή να παρεύουμε στην ε, Λιβύη. Εγώ βέβαια πάντα έλεγα ότι έτσι όπως είχε κατάσταση πριν πάρουμε αυτή την απόφαση, είμαστε σε ένα διέξοδο. Ανάμεσα σε σκύλα και χάρη είτε να παρεύουμε είτε δεν παρεύουμε, ήταν και τα δύο κακά. Τι άλλο όμως θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει. Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να λάβουμε περισσότερο υπόψη μας τη δυσκολία και την πολυπλοκότητα της κατάστασης και να είμαστε πολύ πιο υπομονετικοί σε σχέση με τις καθημερινές εξελίξεις. Πρόεδρος, ναι. Συμφωνώ με τη θέση σας. Πρώτα απ' όλα μια παρατήρηση όσον αφορά τις διαφορετικές προσεγγίσεις. Στη Βοσνία στο πέραν όλων των παραγόντων που διαφέρουν τόσο ή μεταξύ των περιοχών αυτών, εμείς ε, είχαμε εκτελεστική εντολή ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ αυτό δεν συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση, δεν υπάρχει εκτελεστική εντολή στη Λιβύη. Και όπως φαίνεται οι τοπικοί μας συνομιλητές ε, βρίσκονται σε κάπως άναρχη κατάσταση. Και επίσης είναι αρκετά καχύποπτη Ακόμα και όταν πάμε να συζητήσουμε οποιαδήποτε εκτελεστική εντόλη, δεν θέλουν ε, να επηρεάσουμε θέματα τα οποία θέλουν να ιδιοποιηθούν οι ίδιοι. Δεν έχουμε λοιπόν την ικανότητα σήμερα. Εγώ σας ομολογώ μίλησα για ενδιασμούς, προβληματισμούς γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ποια θα ήταν η λύση. Και πάλι συμφωνούμε, και η πλειοψηφία εδώ στο Κοινοβούλιο, ότι έχουμε κάποιο ρόλο να διαδραματίσουμε στο να βοηθήσουμε τη Λιβύη για θέματα ασφαλείας και για θέματα νοικοδόμησης. Ωστόσο, το ερώτημα που τίθεται σήμερα, που θέτω εγώ, σήμερα είναι η παρουσία μας εκεί έχει κάποια χρησιμότητα υπό την παρούσα της μορφή δεδομένων των ελάχιστων αποτελεσμάτων που μπορούμε να ελπίζουμε να επιτύχουμε. Σας ομολογώ, είναι μια ερώτηση που με απασχολεί πολύ και δεν ξέρω ποια θα ήταν η απάντηση. Εγώ έχω αρκετές αμφιβολίες και δεδομένου των όσων ακούω σήμερα και ευχαριστούμε για όλη αυτή την ενημέρωση. Όλα αυτά όσα ακούμε σήμερα εντείνουν τους ενδιασμούς μου. Δυστυχώς φοβάμαι ότι σε κάθε περιοχή κρίσης, διενέξεων, όπου νομιμοποιούμαστε να δράσουμε βρισκόμαστε σε παρόμοιες συνθήκες. Έχουμε αυτές τις αποστολές που ονομάζω εγώ προσφυματικές αποστολές. Είμαστε εκεί γιατί υποτίθεται πρέπει να είμαστε ανεξάρτητα του τι μπορούμε πραγματικά και ουσιαστικά να επιτύχουμε. Κατά την άποψή μου λοιπόν αυτό αποτελεί πρόβλημα. Άννα, παρότι ήρθε στη μέση τη συζήτηση, ίσω θα μπορούσε να μα μοιραστεί μαζί μα τη δική σου εμπειρία από τη Λιβύη, γιατί ήσουν εκεί πρόσφατα. Ανέφερα μόλι τώρα του συνδυασμού μου όσον αφορά την αποστολή εκεί, για την οποία όλοι είχαμε πιέσει να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί εκεί. Θέλαμε να υπάρχει ευρωπαϊκή παρουσία στη Λιβύη, να προσφέρει εργασία στη Λιβύη, αλλά σήμερα δεν πιστώνουμε Δεδομένη τη αβέβαιη κατάσταση, τη άναρχη κατάσταση, διαπιστώνουμε μια αναποτελεσματικότητα όλων αυτών. Και αναρωτιόμαστε κατά πόσο είναι ωφέλιμη η παρουσία αυτή, η δική μα εκεί. Ζητώ που δεν ήρθε νωρίτερα, αλλά μιλούσα στο Λονδίνο με θέματα ασφάλειας του Νότου και η Λιβύη βέβαια ήταν ένα από τα θέματα που θίξαμε. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήμουνα στη Λιβύη και εκεί μάλλον εκεί πήγα στα γραφεία της Γιούμπαμ στους ε, επαγγελματίες εκεί, οι οποίοι με εξέπληξαν πραγματικά με τις προσπάθειες που κάνουν και τον επαγγελματισμό τους. Από την άλλη όμως, οι ίδιοι αναγνωρίζουν τα όρια το... του τι μπορούν να κάνουν. Γιατί εμείς ναι μεν σπέρνουμε κάποιους σπόρους, αλλά δεν ξέρουμε αν κάποιος θα ρίξει νερό για να γίνουν οι σπόροι φυτό στη συνέχεια. Κάπως έτσι μπορώ να το παρουμιάσω. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα διαρθρωμένο. Υπάρχουν δύο δομές, για παράδειγμα, για την θαλάσσια διάσταση. Συνδεδεμένη λοιπόν η αστυνομία για τη θάλασσα με το Υπουργείο Εσωτερικών και οι φύλακες με το Υπουργείο Άμυνας. Αλλά από την άλλη μεριά δεν έχουν εξοπλισμό ή έχουν κάποιον εξοπλισμό αλλά δεν έχουν καθόλου ικανότητες. Είναι δύσκολα τα πράγματα και μας το είπαν οι συνομιλητές μας ότι βεβαίως και είναι πολύ πρόθυμοι οι Λίβοι να μάθουν και να συνεργαστούν με τους δικούς μας δεν ε, τα καταφέρνουν πάντα γιατί δεν βρίσκονται στις θέσεις που θα έπρεπε να βρίσκονται. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι δυνατόν να ασχολούμαστε με θέματα ασφάλεια συνόρων αν δεν έχουμε ασφάλεια. Ε, η ασφάλεια δεν υπάρχει. Αυτή είναι ανύπαρκτη. Δεν υπάρχει ούτε αστυνομία, ούτε πραγματικό στρατός. Τίποτα. Είναι καταστραμμένα. Υπήρχε η ασφάλεια που ήταν ε, μισθοφόρη βέβαια του Πρωθυπουργού. Δεν υπήρχε ασφάλεια τελικά. Είναι μόνο η παραστρατιωτική. Και δεν έγινε τίποτα για να αντιμετωπιστούν αυτές οι βασικές ανάγκες σε ασφάλεια δηλαδή να οργανωθεί κάποια επιχείρηση με κατάρτιση στρατιωτικών δυνάμεων, ε, αφοπλισμού των παραστρατιωτικών ώστε να ενταχθούν στις τακτικές στρατιωτικές δυνάμεις, ε, δεν έγινε. Οπότε τώρα ε, αυτοί οι παραστρατιωτικοί, προφανώς τους οποίους έχουν ενταχθεί από τρομοκράτες μέχρι δεν ξέρω τι, ε, αυτοί εντάσσονται σιγά, σιγά παντού. Οπότε και εγκληματίες και σιγά σιγά διαχέονται παντού. Ακόμα και το θέμα των ναρκωτικών έπεσε όταν ήμουν εκεί σε σχέση με τους παραστατητικούς αυτούς. Άρα τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Κάθε φορά που πάω, ακόμα και όταν πήγαμε αποστολή της Επιτροπής Εξωτερικών από εδώ, είδαμε ότι τα κράτη-μέλη αντιστέκονται προκειμένου να υπάρξει ένα συντονισμό στα πλαίσια τη κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Δεν το θέλουν. Γιατί, Γιατί κάποιε χώρε βέλη σκέφτηκαν ότι αν οι δικοί τους βρεθούν στο Υπουργείο Άμυνα Εσωτερικών κτλ, ίσως να μπορούν έτσι να διασφαλίσουν ότι εκείνοι θα προτιμηθούν για τις προμήθειες στη συνέχεια. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν υπήρχε μεγάλη προθυμία ούτε από την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, ούτε από τα κράτη-μέλη. Και για πρώτη φορά αυτή τη φορά, για πρώτη φορά, επειδή η κατάσταση είναι τόσο άσχημη, εκτός ελέγχου, πραγματικά επικίνδυνη για όλους. Μετά την ε, επίθεση στη ρωσική πρεσβεία, έφυγαν οι Ρώσοι. Επευκαιρία, εγώ πήγα αφού μας είχε πει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ότι θα έκανε ακριβώς αυτή τη δουλειά στη Λιβύη και ήταν πολύ περήφανος. Και όταν ρώτησα στη Λιβύη μου είπανε μα αυτά τα πράγματα του ΝΑΤΟ ναι προετοιμάζονται να γίνουν αλλά δεν γίνονται. Το χαρτί μόνο ετοιμάζεται, υπογραφή ναι. Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να υπάρξει μια συνολική συντονισμένη προσπάθεια για να οικοδομηθούν οι ικανότητες στη χώρα αυτή και η ασφάλεια και ο στρατός. Επίσης μου είπαν, πρέπει να σας το πω και αυτό, ήταν μια σοβαρή πηγή, ότι η Λίβη είναι τόσο απελπισμένοι και ο Πρωθυπουργός Και ενώ μας ζήτησαν ξανά και ξανά ε, μάς το ΝΑΤΟ και δεν είδαν να γίνεται τίποτα. Και όντας πεπισμένος ο Πρωθυπουργό ότι είναι θέμα εξοπλισμού, του το βάλανε ίσως στο μυαλό αυτό, ήταν ε, έτοιμοι να αγοράσουν εξοπλισμό από τους Ρώσους. Οι Ρώσοι τώρα φύγανε, τουλάχιστον για κάποιο διάστημα. Συνεπώς η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Βλέπουμε ότι υπάρχει διάθεση, αλλά η πραγματικότητα είναι πολύ πιο δύσκολη τώρα από ό,τι ήταν πριν από δύο χρόνια. Και εμείς πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αποτύχαμε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω όταν λέμε εικονική, εικονική αποστολή. Εγώ θα έλεγα ότι καλύτερα να πούμε avant-garde αποστολή, δηλαδή πρωτοπόρος, η, η αιχμή της αποστολής. Ε, είχαμε πολύ μεγάλη αποστολή και στο Κωσυφοπαίδιο και μία, ε, ένας, ε, εκτελεστική εντολή μου δεν είναι η λύση. Πρέπει να δείξουμε και πώς πρέπει να γίνονται τα πράγματα στους ε, υπεύθυνου εκεί. Επιτρέψτε μου να σας δώσω μία προοπτική. Ήμασταν όλοι υπερενθουσιασμένοι μετά την πτώση του Καντάφ και όλοι θέλαμε να κάνουμε κάτι, να προσφέρουμε. Ε, ε, εξετά, ήμασταν εκεί το Μάιο φέτος, δηλαδή έξι μήνες περίπου. Ε, εν συνεχεία πρόσφατα διαπιστώσαμε αυτές τις ε, τραγωδίες στη Μεσόγειο που μας πείθουν τους πάντες ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι και εμείς είμαστε στην βέλτιστη θέση να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Έχουμε εμπειρία στην διαχείριση ε, συνόρων, έχουμε επίσης τη δυνατότητα συνεργασίας με εταιρείε παροχής ασφα... υπηρεσιών ασφαλείας, άμα δεν μπορούμε εμείς να το κάνουμε. Και εν πάση περιπτώσει πρέπει να κάνουμε μία προσπάθεια και να δείξουμε ότι ε, είμαστε αποφασισμένοι να πράξουμε κάτι. Δεν είναι δυνατόν όλες αυτές οι αποστολές να σημειώσουν επιτυχία, να είναι ε, επιτυχημένες. Ε, Πρέπει να... Οι αποφάσεις λαμβάνονται από τους πολιτικούς, από τα πολιτικά αφεντικά μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αν μου επιτρέπετε, εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αυτά. Ο Πρόεδρος. Ωραία, λοιπόν, ευχαριστούμε. Δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητές που θα ήθελα να το λόγο. Κλείνω εδώ λοιπόν τη συζήτηση για την ε, Γιουμπαμ Λιβύη. Ευχαριστώ τον κύριο που ήρθε εδώ και να μας κάνει την ενημερωσή του. Είναι ένα θέμα φυσικά για το οποίο θα μένουμε σε επαφή και ελπίζω ότι στην επόμενη επίσκεψή του στην Ευρώπη θα μπορούσαμε να υποδεχθούμε εδώ τον αρχηγό της Αποστολής. Ελπίζω να μην χρειαστεί να μείνει μόνιμα αποσπασμένο στην Τρίπολη και να μπορέσει λιγάκι να ταξιδέψει. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα θέμα που μας απασχολεί ιδιαίτερα και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να το ξανασυζητήσουμε. Μην διστάσετε λοιπόν να μας παράσχετε οποιαδήποτε νέα στοιχεία που μπορεί να χρειάζεται να συζητήσουμε και η Άννα παρακολουθεί την κατάσταση ούτως ή άλλως. Θα συζητήσουμε λοιπόν τις όποιες νέες εξελίξεις. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Θα περάσω την Προεδρία στον Αντιπρόεδρο Παλέτσκης, ο οποίος θα με αντικαταστήσει. Σας ευχαριστώ. <laughs> Dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να συνεχίσουμε με τις συζητήσεις μας. Θα συζητήσουμε τώρα την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφαλείας και άμυνας. Καθώς γνωρίζω, πολλές ήταν οι τροποποιήσεις, πάνω από 150 και οι περισσότερες από αυτές κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση υποστηρίζονται από όλες τις μεγάλες πολιτικές ομάδες. Η ψηφοφορία λοιπόν στην ΑΦΕΤ ε, δεν θα λάβει χώρα αυτή την εβδομάδα όπως σχεδιαστεί. Θα λάβει χώρα στην Σύνοδο του Στρασβουργού. Καλό τώρα την κυρία Κοπά να μας πει δύο λόγια για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας όλους όσοι συνέβαλαν στην ε, σύνταξη αυτής της έκθεσης και ειδικότερα τους κοιόδης συζητητές για την άριστη συνεργασία τους. Η έκθεση αυτή αφορά τη συζήτηση για το πώς θα εκπληρώσει τις προσδοκίες όσον αφορά τις υποχρεώσεις ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύο μήνες πριν το, η συνάντηση του Συμβουλίου το Δεκέμβριο Θα αφορά λοιπόν το εξέταση των ζητημάτων άμυνας. Για μένα αυτή η έκθεση, όπως ανέφερα ήδη, θα πρέπει να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα από το Κοινοβούλιο στο Συμβούλιο. Όπως είπατε, 150 ήταν οι τροπολογίες και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που τις υπέβαλαν. Το 1 τρίτο σχεδόν των υποβληθισών ε, τροπολογιών συμπεριλαμβάνονται στι 12 συμβιβαστικέ τροπολογίε που συζητήσαμε την περασμένη εβδομάδα την Δετάρτη, την Δετάρτη στο Στρασβουργό με τους γεωδησίτες. Μια τελευταία μορφή συμβιβαστική τη έκθεση που οριστικοποιήθηκε σήμερα εστάλει στου Κιώδης δύο ώρε περίπου πριν τη συνάντησή μα. Πείτε μου παρακαλώ αν είστε ικανοποιημένοι με αυτούς τους συμβιβασμούς ε, Διαφορετικά θα ψηφίσουμε τις εν λόγω παραγράφου ξεχωριστά. Πρώτα απ' όλα λοιπόν μερικές παρατηρήσεις επειδή θα δείτε τις συμβιβαστικές τροπολογίες ε, έχετε την γνωμοδότηση και νομίζω ότι η συζήτηση, το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης έχει ήδη γίνει. Πρώτο σημείο λοιπόν. Κατά τη σύνταξη αυτή τη έκθεση, ε, ήμουν κατά και είμαι ακόμα κατά του να κάνουμε αναφορά σε συγκεκριμένε χώρε ή περιοχέ δεν πρέπει να μετατρέψουμε αυτή την εκθέση σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο και να πούμε τα πάντα. Ευχαριστώ τους κοιόδης που δέχτηκαν αυτή την αρχή και δεν κατονομάζουν συγκεκριμένες χώρες και περιοχές. Αυτή είναι η αρχή την οποία θα ακολουθήσω και εγώ κατά τη λίστα ψηφοφοριών. Δεύτερο σημείο. Το επιχειρησιακά κεντρικά στρατηγία. Ξέρω ότι είναι σημαντικό ζήτημα για πολλούς συναδέλφου λόγω των εθνικών τους θέσεων. Έχω μια τροπολογία από τον κύριο Ντάνζαν, όπου ακόμα και η αναφορά μιας ε, οργανωτικής κυψέλη ε, για τις επιχειρήσεις τον ενοχλεί και θέλει να τη διαγράψει. Η ιδέα αυτή μιας επιχειρησιακής κυψέλης βασίζεται σε αυτά που άκουσα εγώ από τους επικαφαλής αποστολών και στρατιωτικών αποστολών. Μου λένε ότι όταν έχουν να αντιμετωπίσουν στρατιωτικά ζητήματα επιτόπου χωρίς να αναφέρονται στις Βρυξέλλες και να ζητούν γνώμη για κάθε διοικητική λεπτομέρεια. Είναι ένας τρόπος αυτός Εντάξει, ας μην μιλήσουμε για επιχειρησιακό στρατηγείο, δηλαδή είναι δύσκολο, είναι η θέση του Κοινοβουλίου, γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται να περάσει, αλλά τουλάχιστον μία οργανωτική δομή ε, Κυψέλη, συγγνώμη, είναι απαραίτητη, πιστεύω. Και θα στείλω ένα email στην Κρυτανζά, αλλά μπορούμε να το δούμε μαζί. Πιστεύω ότι καλό θα ήταν να μην επιμείνουμε σε αυτό. Τρίτο σημείο. Έλαβα δύο τροπολογίες από τους πρασίνους, δυστυχώς δεν βρίσκεται εδώ κανένας από τους πράσινους, που αφορούν μια παρανόηση κατά την απόψή μου που είχαν αυτοί όσον αφορά το ρόλο της ΚΕΠΑ στα εξωτερικά σύνορα. Μιλάμε για τι τροπολογίες 31 και 33. Εγώ ποτέ δεν είπα στην έκθεση ότι η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνα έχει να παίξει ένα ρόλο σύμφωνα με τις συνθήκες ε, για να επιλαμβάνεται των εξωτερικών συνόρων. Λόγω μια παρανόηση θεωρούν ότι είναι απαραίτητο να επιμείνουμε δι ότι αυτό δεν είναι δουλειά τη κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνα. Εγώ το γνωρίζω. Δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου. Και θα ήθελα τουλάχιστον η γραμματεία του να το σημείωσε και να περάσει το μήνυμα αυτό ότι θα προσπαθήσω να δεχτώ ένα κομμάτι της δικής τους τροπολογίας αλλά το να επιμένουμε για κάτι που δεν έχω πει δεν μπορώ να το δεχτώ θα προσπαθήσω να κάνουμε κατά τμήματα ψηφοφόρια τουλάχιστον για τα κάποια σημεία των τροπολογιών τους που μπορώ να δεχτώ τέταρτο σημείο στην τροπολογία 110 ο κύριος Νταφ ε, θεωρεί απαραίτητο να προσθεθεί κάτι το ευρύτερο πεδίο επιχειρήσεων όπου λέει ειδικότερα στη γειτονική περιοχή, αυτό προσθέτει, ειδικότερα στη γειτονική της περιοχή, αυτό μπορεί να γίνει κατανοητό με δύο τρόπους. Μπορεί να περιορίζουμε τις φιλοδοξίες, το οποίο μπορεί να είναι σωστό και να μπορούμε να το δεχτούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παρέχει ασφάλεια σε όλο τον κόσμο. Αυτό ξεπερνά κατά πολύ τις δυνατότητες μας, ειδικότερα σε εποχές κρίσης. Με αυτό το σκεπτικό μπορώ να το δεχτώ. Αλλά θα μπορούσαμε να καταλάβουμε και αλλιώ αυτή την τροπολογία. Ειδικότερα στην περιοχή ότι έχουμε υποχρέωση να δράμε με επιχειρήσει στην περιοχή μα. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι, για παράδειγμα, στο Νότιο Κάφκασο, έχουμε υποχρέωση να παρέμβουμε. Δεν είναι σαφέ αυτό που προτείνεται. Γι' αυτό θα ήθελα να το συζητήσουμε κάπως οι δυο μα, για να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση που θα καταστήσει το κείμενο πιο σαφέ από ό,τι είναι. Μπορούμε λοιπόν διμερώς να το εξετάσουμε και το τελευταίο που είχα να πω. Α, το απευθύνω κυρίως προς την Κομισιόν. Το ΕΛΚ πολύ σωστά υπέβαλε τροπολογίες που αφορούν την ενδιάμεση εκθέση της ε, κυρίας Άστον. Η ενδιάμεση έκθεση πρέπει να είναι αυτό που λέει το όνομά της, μια προσωρινή έκθεση. Κατά με είναι σημαντικό να συμπεριλάβουμε στο κείμενο κάτι σημαντικότερο από μια αναφορά σε μια ενδιάμεση έκθεση. Και η ερώτηση προ την Κομισιόν είναι μπορούμε να δεχτούμε στο μέλλον να αναφέρουμε την τελική έκθεση της Λεδισάστον. Να ευχαριστήσω όλους που συνεργάστηκαν μαζί μου. Δημερώς να συζητήσουμε για τα σημεία που μας απασχολούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία σας και την ε, μεγάλη σας διάθεση συνεργασία κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μας. Ευχαριστούμε πολύ. Από ό,τι καταλαβαίνουμε υπάρχουν κάποια σημεία που είναι επίμαχα. Οπότε οι σκιώδες συζητητέ και πρώτα απ' όλα ο κύριος Γκάλερ. Μια που ο πρόεδρός μας δεν είναι εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους του κύριου Ντανζό θα ήθελα αλλά και εκ μέρου και εμού του ιδίου. Ε. Θέλω να σα συγχαρώ για την έκθεση αυτή, που πιστεύω ότι στέλνει ένα πραγματικά ισχυρό πολιτικό μήνυμα προ του αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων. Αν εφαρμοσόντουσαν αυτά, τότε θα είχαμε πράγματι μια πιο ισχυρή κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Ο κύριος Τανζάν είναι πολύ ευχαριστημένος από την συνεργασία Τώρα έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Αναφερθήκατε σε ποια για την 70? Μικρόφωνο παρακαλώ, μικρόφωνο. Κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη όσων βρίσκονται επί τόπου, χρειάζεται, δεν ξέρω αν θα βρούμε κάποια συμφωνία, λάβετε το υπόψη σας. Μα στους Κιώδης συζητήθηκε. Ο κύριος Στενζό δεν το έθεσε στη συνεδρίαση, αλλά είδα τις τροπολογίες. Ίσως μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτό αργότερα. Πρόεδρος, ναι, μήπως διμερός να το δείτε. Για το υπόλοιπο δεν έχω πρόβλημα, μόνο για το θέμα αυτό της ε, επίσημης, του επίσημου οργανωτικού πυρήνα. Η Κυψέλη, οργανωτική μονάδα. Εντάξει, θα το δείτε αυτό. Οι υπόλοιποι. Τελειώσατε. Ωραία. Η κυρία Νίτς τότε, εκ μέρους του Άλντε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να συγχαρώ την συνάδελφο Κοπά για την εξαίρετη έκθεση. Και ευχαριστώ πολύ και για την εξαίρετη συνεργασία που είχαμε μεταξύ μας. Είμαι σκιώδη συζητήτρια για την έκθεση αυτή και εκτιμώ ιδιαίτερα την προσπάθεια που κάνατε προκειμένου να συντάξετε συμβαστικές τροπολογίες οι οποίες να λαμβάνουν υπόψη πολλές από τις δικές μας τροπολογίες. Και παρόλα αυτά η έκθεση παραμένει με συνοχή και ευθυγραμμίζεται στο συνολικό κλίμα. Οπότε σας ευχαριστώ για αυτό. Τώρα όσον αφορά την τροπολογία DAF. Εννοείται ότι πρέπει να το συζητήσετε και μαζί του, αλλά νομίζω ότι ξέρω τι εννοεί. Γιατί είναι πολιτική της άλλη αυτή. Εμείς πιστεύουμε ότι Έχουμε καταρχήν αρμοδιότητα και ευθύνη για την γειτονική μας περιοχή. Με την έννοια δηλαδή το ότι αν εμείς δεν λάβουμε υπόψη μας και δεν ασχοληθούμε με την, γείτονα, την γειτονική μας περιοχή, τότε ποιος θα το κάνει. Αυτό είναι το πνεύμα της τροπολογίας DAF. Όχι ότι πρέπει να παρεμβαίνουμε κάθε φορά και οποτεδήποτε κάτι συμβαίνει στην γειτονική περιοχή, αλλά το πνεύμα είναι ότι αν εμεί δεν ασχοληθούμε με τη δικιά μα γειτονική περιοχή, ε, ποιος άλλος θα το κάνει τότε. Συνεπώ ίσω μπορείτε να προσπαθήσετε να βρείτε μια διατύπωση με την οποία να συμφωνείτε και δύο, αλλά είμαι περίπου σίγουρη ότι αυτό εννοούσε, γιατί αυτή είναι η δικιά μα γραμμή, βλέπετε, στην άλλη με την οποία όλοι συμφωνούμε εδώ και καιρό. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Άλλος. Ποιος άλλος θέλει να σχολιάσει. Ο κύριος Μπαϊτικόφερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μιλώ εκ μέρους του συνδέλφους μου κ. Κρόνμπερκ, ο οποίος ταξιδε... δεν μπόρεσε να είναι παρόν και είναι σκιώδης εισηγητής, είχε προβλήματα στην μετάβαση. Καταρχάς είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και με τη δομή και με το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου της ε, γνωμοδότησης και ευχαριστούμε την εισηγήτρια που ενσωμάτωσε πολλές από τις τροπολογίες μας. Έχω δύο σχόλια. Το ένα αφορά ε, στα εξωτερικά σύνορα. Ε, και Ζητώ συγγνώμη ε, που δεν ήμουν παρόν προηγουμένως, αλλά έπρεπε να ψηφίσουμε στην Ήτρε. Γι' αυτό θα είμαι σύντομος. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Πιστεύουμε ότι η προστασία των συνόρων δεν είναι ε, μία πτυχή, ένα στοιχείο της ε, κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Δεύτερον, το θέμα προϋπολογισμών και δυναμικού δυνατοτήτων. Δεν πιστεύω ότι η έλλειψη δυνατοτήτων οφείλεται στην έλλειψη προ... προϋπολογισμών. Διότι αν ε, ακόμα και όταν η χρηματοδότηση ήταν καλύτερη, πάλι είχαμε προβλήματα ικανοτήτων. Τα, πιστεύω ότι έχουμε μείωση των ικανοτήτων μας επειδή δεν συνεργαζόμαστε όσο θα έπρεπε. Θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας και τις προτεραιότητες μας σαφέστατα προς αυτή την κατεύθυνση και γι' αυτό θέλω να τονίσω ότι η έκθεση Galler είναι πολύ συγκεκριμένη και πολύ σαφής σε, αυτό, σε αυτή την πτυχή. Τονίζει ότι πρέπει να συνεργαστούμε ε, και ότι θα πρέπει να συγκεράσουμε τις, ε, τις, τις απόψεις μας, τη συνεργασία μας στις διάφορες πλευρές ε, για να βελτιώσουμε τις ικανότητές μας. Και αυτό είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Η συνεργασία πρέπει να ενισχυθεί και το ε, υπερβολικό, το πλεονάζον δυναμικό στον τομέα αυτό θα πρέπει να μειωθεί. Κύριε Κοπά, ευχαριστώ. Συμφωνώ μαζί σας και αν μπορείτε να αναφέρετε ποιες είναι οι πιο σημαντικές τροπολογίες σε αυτό το ειδικά το σημείο που είπατε. Ε, παρακαλώ, διαβάστε την παράγραφο 8. Δεν νομίζω ότι... αναφέρω εδώ ότι ο στόχος της ΚΠΑ είναι να περιλάβει και τα εξωτερικά σύνορα. Αναφέρω και αυτό αυτούς που έχουν σχέση ή άπτονται των εξωτερικών σύνορων, που αφορούν τα εξωτερικά σύνορα. Είναι στην παράγραφο 8, δεν λέω ποτέ και τα εξωτερικά σύνορα. Περιλαμβανομένων και αυτών που αφορούν τα εξωτερικά σύνορα λοιπόν. Βάσει το άρθρο 21 δεν είναι στην συνθήκη τα εξωτερικά σύνορα. Λοιπόν, καταστατικού του εθνών του και στόχους του χάρτη του Παρισιού, περιλαμβανομένου και αυτών που αφορούν τα εξωτερικά σύνορα. Ενώ ότι όλοι αυτοί οι στόχοι αφορούν την, τον, ε, έχουν τον ίδιο σκοπό να αυξήσουν τις ικανότητές μας. Αν μπορείτε να δεχτείτε αυτή την παράγραφο, την 8, θα μπορέσω εγώ να δεχτώ και το δεύτερο μέρος της τροπολογίας, μας, ε, της τροπολογίας σας από τη λέξη record στη λέξη stabilization. Ωραία, θα τα πούμε διμερώς. Ε, ο πρόεδρος, ε, η τελική έκδοση της γνωμοδότησης έχει υποβληθεί στον κύριο Ντανζόν και θα δοθεί και σε όλα τα μέλη της ΕΔΕ τελική έκδοση. Μπορούμε τώρα να συνεχίσουμε με το επόμενο θέμα που είναι η τεχνολογική και βιομηχανική βάση της Ευρωπαϊκής Άμυνας του κυρίου Γκάλερ. Ευχαριστώ. Είχαμε, αν θυμόσαστε συνάδελφοι, αυτή την αξίση που βασίζεται στο άρθρο 50 και την είχαμε επεξεργαστεί μαζί με την Ήτρε. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι πρέπει να εκτιμήσω θετικά ότι από τη μία πλευρά έχουμε μία μεγάλη απικάλυψη στους τομείς αλλά και μία πολύ μεγάλη σύγκληση απόψεων. Αυτό δεν με ανησυχεί τόσο πολύ. Αυτό που με ανησυχεί εμένα είναι ότι δεν θέλω να, ότι θέλω να αποφύγω επαναλήψεις. Σας είπα ότι θέλω να καταλήξω στις στην καλύτερη ουσία συγκεράζοντας τις δύο εξέσεις. Είχα συντάξει 10 συμβιβαστικέ τροπολογίες και είχαμε και μία συνάντηση των σκιωδών την περασμένη εβδομάδα που δεν είχε αρκετή συμμετοχή ως συνέπεια αυτού σας ε, παρακαλώ ε, προσέξτε δύο, θα κάνω δύο παρατηρήσεις για να έχουμε και τη συνεργασία των πρασίνων. Γίνονται πολλαπλές αναφορές ε, στον τομέα της απασχόλησης, στη βιομηχανία και στη συμβιβαστική ένα θέλω λίγο να αμβλύνω την εστίαση στις, ε, στις θέσεις εργασίας. Εμείς έχουμε την ΚΠΑ διότι αντιμετωπίζουμε προκλήσεις και απειλές και χρειαζόμαστε μια ισχυρή βιομηχανική βάση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απειλές και προκλήσεις. Συνεπώς, ε, με το θέμα αυτό συνδέονται και ορισμένες θέσεις εργασίας. Αλλά δεν Νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος για μια ισχυρή κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, δηλαδή ο εργασιακός τομέας. Ε, ε, ε, εάν μας αναθέσουν έργα οι Ρώσοι ή οι Κινέζοι, εντάξει, θα έχουμε περισσότερες θέσεις εργασίας, αλλά αυτό είναι μια παράπλευρη επίπτωση του τομέα. Ένα άλλο σημείο αυτό είναι ένα ε, σημείο που δέχτηκα να διαγράψω και επίσης για να κάπως ικανοποιήσω τους συναδέλφους τους πράσινους ε, θα ήθελα να, να αναφέρω και το θέμα του τηλεχειρισμού των αερο, τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών θα προσθέσω τη λέξη SAM, μερικά, μερικά, ορισμένα αν θέλετε. Αυτά ήταν τα δύο σημεία. Uh, the uh... αυτά ήταν οι δύο παρατηρήσεις. Κατά τα άλλα πιστεύω ότι υπάρχει μια ευρεία συνενετική βάση και δεν προβλέπω να δημιουργηθούν προβλήματα, να προκύψουν προβλήματα ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Εάν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, ο κύριος Βίτεκοφερ, στην περίπτωση αυτή είμαι όντως ο σκιώδης εισηγητής Όντως, λέει ο πρόεδρος, είσαστε. Μου δώσατε το λόγο ήδη, αλλά τώρα θα επανέλθουμε με το καπέλο του σκιώδου συζητητή. Πρόεδρε, θέλω να πω ότι καλωσορίζουμε αυτή την έκθεση και είμαστε και ευτυχείς με το αποτέλεσμα της ε, συνάντησης των σκιωδών συγητών την περασμένη εβδομάδα τα αποτελέσματα τα διαβιβάσαμε σε όλους σας. Είναι πολύ σημαντικό στην παράγραφο 3 του σχέδιου έξεσης να δώσουμε ένα σαφέστατο μήνυμα ότι ορισμένες από αυτές τις εξαγωγές τεχνογνωσίες και τεχνολογίες από πλευράς ασφάλειας μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ευρώπης. Πρέπει να πω ότι αυτό το θέμα δεν έχει ξεκαθαριστεί ποτέ και νομίζω ότι αυτό είναι ευκαιρία να το κάνουμε σε αυτή την έκθεση. Επίσης στην παράγραφο 8, 5, 17 που εστιάζονται τα προβλήματα του κατακαιρματισμού, της επανάληψης και του πλενάζοντος δυναμικού ή δίνουν ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Ένα συγκεκριμένο θέμα θέλω να θίξω είναι η τροπολογία 59 η οποία έχει κυρίως σχέση με τη Ρουμανία. Η Ρουμανία θέλει να αγοράσει 12 ε, μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16. Από ό,τι φαίνεται η Ρουμανία δεν έχει προκηρύξει ένα δημόσιο διαγωνισμό, ούτε έχει κοιτάξει άλλες εναλλακτικές λύσεις όπως το Eurofighter και άλλα μαχητικά αεροσκάφη. Κατά τη γνώμη μας αυτή η διαδικασία είναι μία παρατυπία και παραβιάση του κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία τέτοια συμφωνία θα, αποδυ... θα αποδυναμώσει, ε, θα εξασταμιώσει ε, την ε, ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας αεροπορική αεροπορικού δυναμικού. Γι' αυτό θα ήθελα στην τροπολογία 59 να γίνει μία σαφής ε, αναφορά στις ρουμανικές αρχές, ιδίως επειδή αυτό συνάδει και με την πολιτική της Κροατίας ε, και της Σλοβακίας που ενδεχομένως να συνάψουν παρόμοιες συμφωνίες ε, προμήθειας. Είναι λοιπόν μία, ένα σημείο που ο κύριος Γκάλερ προς το παρόν θα μπορέσει να δείξει και να τονίσει ότι η ευρωπαϊκή αμυντική έρευνα δεν θα πρέπει να χρωματοδοτείται από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Θα πρέπει να πείσουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν πιο ε, καλή χρήση του προϋπολογισμού τους, τουλάχιστον της πτυχής εκείνης που, μέσω της οποίας χρηματοδοτούν τη στρατιωτική τους άμυνα. Πρέπει να πιέσουμε τις, τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Εφόσον έχουμε περιορισμένο ερευνητικό budget, ε, το οποίο ήδη μας δένει τα χέρια, είναι πολύ περιοριστικό, εάν διευρύνουμε τη δυνατότητα χρηματοδότησης ε, βιομηχανικού και και βιομηχανικής και στρατιωτικής τεχνολογικής έρευνας θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο η πίεση. Ε, εδώ διαφωνώ με την ε, στρατηγική, με την προσέγγιση. Ξέρω ότι έχει ψηφιστεί σε άλλες εκθέσεις, αλλά δεν θα ήθελα να υπάρχει εδώ. Ο Πρόεδρος, η κυρία Κοπά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Μακλεγκαλέρ για αυτή την έκθεση. Δεν είμαι σκιώδη, αλλά την παρακολούθησα στενά ω συντονιστρία των σοσιαλιστών. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη γιατί με αυτέ τι δύο εκθέσει ε, θα στείλει το Κοινοβούλιο ένα ισχυρό μήνυμα. Είναι συμπληρωματικέ αυτέ οι εκθέσει, καλύπτουν διαφορετικέ πτυχέ και πιστεύω ότι στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου όπου ελπίζουμε να ψηφιστούν το μήνυμα προς το Συμβούλιο θα είναι ιδιαίτερα ισχυρό. Συγχαρητήρια και πάλι και ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας σε όλη τη διαδικασία σύνταξη αυτών των διεκθέσεων. Ευχαριστούμε. Ο Πρόεδρος. Η κυρία Σίλβια Χάινς Χούμπερ πρέπει να είναι εδώ και Κομισιόν. Ε, ναι, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα είμαι πολύ σύντομη. Εμείς στην Κομισιόν γενικά καλωσορίζουμε ιδιαίτερο σε αυτή την έκθεση να συμφωνήσω με τα όπα. Όσα είπε η κυρία Κόπα, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την έκθεση. Πολλές συγκεκριμένες ε, ιδέες και ακριβείς που εκφράζονται και στην ανακοίνωση της Κομισιόν υπάρχουν σε αυτή την έκθεση, γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες ε, και χαιρόμαστε που έχουμε την υποστήριξη του Κοινοβουλίου σε αυτές τις ιδέες που εκφράστηκαν στην ανακοίνωση τη Επιτροπή. Ευχαριστούμε πολύ, ε, Πρόεδρο Ευχαριστούμε. Κύριε Γκάλερ, έχετε σχόλια ναι, για την τροπολογία 59 που αφορά τα F-16. Συμφωνώ. Θα τη λάβω υπόψη μου λοιπόν. και όσον αφορά το χαρακτήρα του άλλου προγράμματος η έρευνα και νομίζω ότι στο άρθρο 173 της συνθήκης είναι σαφές ότι αναφέρεται και στο γεγονός ε, ότι και η έρευνα συμβάλλει στη βελτίωση άλλων πολιτικών που επιδιώκουμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έρευνα λοιπόν είναι μια πτυχή που αποτυπώνεται και στις συνθήκες ως επηρεάζουσα και άλλες πολιτικές. Μπορούμε λοιπόν να υποστηρίξουμε βάσιμα ένα χαρακτήρα όχι αποκλειστικά με στρατιωτικό και η πρόταση χρηματοδότησης του προσωπικού όχι μόνο από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι για να βοηθήσει τα κρατημέλη που ισχυρίζονται ότι δεν θέλουν να συνεχίσουν τη χρηματοδότηση. Αυτό μπορεί να διευκολύνει και την επίτευξη των διαφόρων ε, επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ναι, κανείς άλλος. Ωραία, ευχαριστούμε. Καλό λοιπόν τον κύριο Γκάλερ που είναι... Έχει πολλά πράγματα να κάνει σήμερα, να μας μιλήσει για το επόμενο σημείο είναι το σχέδιο γνωμοδότησης για το πρόγραμμα υποστήριξη για την Επιτρήση και παρακολούθηση του διαστήματος. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Τι έχουμε εδώ. Αυτή η γνωμοδότηση αφορά ένα νομοθετικό σχέδιο το σχέδιο γνωμοδότησης λοιπόν έχει τη μορφή τροπολογιών για το προτινόμενο νομοθετικό κείμενο. Οι τέσσερις κατευθυντήριες αρχές για τη δική μας γνωμοδότηση για την Επιτροπή της Ουσίας στην ε, Ήτρε όσον αφορά αυτή τη δήλωση του, για το πρόγραμμα επιτήρησης ε, και παρακολούθησης του διαστήματος οι κατευθυντήρες αρχές είναι ότι αφενός θέλουμε να επισημάνουμε τις επιπτώσεις για τις εξωτερικές υποθέσεις και τις υποθέσεις ασφαλείας και να γίνει έκκληση για νομική βάση για διεθνή συνεργασία. Να καταστεί σαφές ε, ότι οι υπηρεσίες αυτές έχουν και μη στρατιωτική και στρατιωτική φύση. Αυτές είναι οι τέσσερις κύριες κατευθυντήρες αρχές και στην τροπολογία σε μια τροπολογία έχω προτείνει ανεπαναδιατύπωση απλά για να είναι πιο σωστή είναι η τροπολογία 10 η πρόταση τη Επιτροπή λέει κατοχή εισιτήριων εσεστή και επαρκών τεχνικών και ανθρωπινών πόρων για τη λειτουργία του ή ικανοτήτων επεξεργασία δεδομένων. Ε, εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να λέει κατοχή αισθητήρων SST ή δυνατοτήτων επεξεργασίας δεδομένων SST και επαρκών τεχνικών και ανθρωπινών πόρων για τη λειτουργία τους. Αυτή είναι η σωστή διατύπωση, πιστεύω. Κατά τα άλλα, καθώς το βλέπω εγώ, είναι ένα ζήτημα για το οποίο υπάρχει ομοφωνία σε μεγάλο βαθμό. Ευχαριστούμε. Πρόεδρος, θα ήθελα κάποιος να σχολιάσει. Πρέπει τόντως ως και ηγητής των σοσιαλιστών επί του θέματος υποστηρίζω την προσέγγισή σας, κύριε Γκάλερ. Αν δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο, ναι, παρακαλώ. Δεν θέλω να σχολιάσω, αλλά επειδή συμμετέχω στην Επιτροπή Ήτρα για το συντονισμό αυτού του θέματος, νομίζω ότι η αναφορά αυτή στη μη στρατιωτική και στρατιωτική φύση όλων αυτών είναι σημαντική, γιατί στο παρόν σχέδιο της Επιτροπής ΙΤΡΕ αναφέρεται μόνο στην μη στρατιωτική πτυχή. Που δεν είναι κάτι λογικό. Διότι υπάρχουν και μη στρατιωτικά και στρατιωτικά μέσα και θέλουμε συνεργασία και για τα δύο. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι σημαντικό αυτό το σχόλιο και θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους ε, στην Επιτροπή Βιομηχανίας να βοηθήσουμε να το προωθήσουμε αυτό γιατί διαφορετικά νομίζω ότι το σχέδιο κειμένου στην Ήτρε δεν έχει νόημα. Κύριε Μπουτικόφερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να μιλήσω εκ μέρου του σκιώδου συναδέλφου μου του κύριου Γκρόνπακ. Συμφωνώ με τον κύριο Έλλερ ότι πρέπει να προσεγγίσουμε το ζήτημα μη ιδεολογικά. Αλλά εγώ καταλήγω στο αντίθετο συμπέρασμα προσπαθώ να μάθω από αυτά που μαθαίνω ότι γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τι κάνουν με τα διαστημικά απόβλητα. Επειδή το ζήτημα είναι μη στρατιωτικό εκεί, η μη στρατιωτική πλευρά, η αστική πλευρά αναλαμβάνει την ευθύνη. Δηλαδή κινούνται προς ακριβώς την αντίθετη κατεύθυνση. Εγώ δεν είμαι βέβαιος κατά πόσο θα έπρεπε εμείς να επαναλάβουμε την αρχική τους κίνηση και μετά από δύο χρόνια να επανέλθουμε σε αυτό που έκαναν αυτοί μετά από τα όσα έμαθαν και μας έχουν ήδη αποδείξει. Πιστεύω ότι είναι μη στρατιωτικό το ζήτημα αυτό και γι' αυτό το λόγο Ευρω... ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας δεν θα πρέπει να συμμετάσχει. Ευθύνη για αυτό θα πρέπει να έχει η ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος. Ευχαριστώ. Βλέπω ότι εδώ υπάρχουν επίμαχα ζητήματα. Κύριε Γκάλερ. Ίσως καλύτερα πρώτα κύριο Σέιλερ και μετά εγώ στο τέλος. Ναι, νομίζω ότι η ιδέα δεν είναι να στρατιοκοπήσουμε το θέμα. Απλώς ότι υπάρχουν στρατιωτικοί δορυφόροι και αυτό είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. γιατί αν η μη στρατιωτική πλευρά καταστρέψει με ροκέτα έναν δορυφόρο, όπως έγινε με τους Ρώσους και τους Κινέζους, το σύστημα δεν πρέπει να ασχολείται με στρατιωτικά ζητήματα, αλλά να λάβει υπόψη του και τη στρατιωτική πτυχή, γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα αφού υπάρχει και αυτή. Και το γεγονός ότι ο οργανισμός αυτός στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι στη μη στρατιωτική πλευρά, δεν σημαίνει ότι δεν ασχολείται με στρατιωτικούς ε, δορυφόρους, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, γιατί το κοινό δεν τα γνωρίζει αυτά. Συνεπώς, μην ιδεολογικοποιούμε το θέμα και ας καταλήξουμε στην απλή λύση που είναι η πιο πρακτική. Η ιδέα δεν είναι να στατιωτικοποιήσουμε το θέμα, αλλά πρέπει να συνδυάσουμε πληροφορίες, αλλιώς δεν έχει νόημα. Άλλα σχόλια, κύριε Γκάλερ. Θα ήθελα να τελειώσει αυτή η περίεργη παράδοξη κατάσταση όπου δύο Γερμανοί ευρωβουλευτές μιλούν συνεχώς στα αγγλικά. Λοιπόν, μιλώ τη μητρική μου γλώσσα. Ωραία, σωστά όλα ελέγχθησαν, αλλά η οργάνωση δεν γίνεται μόνο από στρατιωτικού, αλλά και από μη στρατιωτικέ δυνάμει. Οπότε από πρακτική απόψεω, όταν όλοι αυτοί λαμβάνουμε υπόψη όλου αυτού του παλιού δορυφόρου και τι δορυφορικέ εγκαταστάσει, δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε ε, αν είναι στρατιωτική ή μη στρατιωτική χρήση. Πρέπει όλου να του καλύψουμε. Πάση φύσεω. Ακριβώ. Ε, άρα μπορεί να, να λειτουργεί ο δορυφόρος για στρατιωτικούς σκοπούς αλλά όχι για στρατιωτικές επιχειρήσεις. Έτσι το βλέπω εγώ ρεαλιστικά. Άρα εξυπηρετεί στρατιωτικούς σκοπούς. Διότι ο θεωρητικός τομέας δεν μπόρεσε να τον ε, καλύψει το δορυφόρο αυτόν. Άρα εξυπηρετεί και συμφέροντα. Είναι λοιπόν μια διαφορετική βάση από την οποία εγώ ξεκινάω. Ο πρόεδρος, βλέπω τη συζήτηση μεταξύ τριών Γερμανών Ευρωβουλευτών μπορεί να κρατήσει πολλή ώρα. Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Εγώ δεν έκανα, δεν επέκρινα τη στατιωτική πτυχή. Απλώς ήθελα να παραμείνω ρεαλιστή, μια ρεαλιστική προσέγγιση. Στην ε, κύριε Γκάλερ, έτσι όπως περιγράψατε τα θέματα, δεν βλέπω καμία αντίρρηση. Είναι να, ε, να, να μπορέσουμε να συλλάβουμε και να διαχειριστούμε όλα αυτά τα διαστημικά σκουπίδια ή τα διαστημικά υπολείμματα τα οποία περιστρέφονται και υπάρχουν. Η γνώση της κατάστασης είναι μία πτυχή. Αλλά η απομάκρυνση αυτών των πολυμάτων είναι και μη στρατιωτική επιχείρηση, έτσι δεν είναι όχι μόνο στρατιωτική. Ε, το θέμα είναι ότι δεν μας ε, αφορά τόσο από πού προέρχεται, ποια είναι η προέλευση των υπολοιμάτων, αλλά πώς θα μπορέσουμε να τα συμμαζέψουμε. Το θέμα είναι θα παίξει, πρέπει να παίξει ρόλο και η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία κατά τη γνώμη μου διόλου δεν έχει καμία αρμοδιότητα σε αυτό το τομέα. Ο πρόεδρος. Α, όχι, ο κύριος Γκάλερ. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε περαιτέρω το θέμα. Α, λοιπόν, λέει ο πρόεδρος, τι επισημείτε. Τα ήταν λοιπόν πολύ επιτυχημένη αυτή η γερμανογερμανική διαβούλευση μεταξύ των τριών σας. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας και λύεται η συνεδρίαση. Η επόμενη συνεδρίαση είναι στις 5 Νοεμβρίου 9.30 το πρωί. Ευχαριστώ πολύ.